Good evening, colleagues. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Σας παρακαλώ όλους να καθίσετε. Για να αρχίσουμε εγκαίρως, είναι πάρα πολύ αυστηρό το χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει και να το τηρήσουμε. Καθίστε παρακαλώ και συζητήσεις εκτός της αιθούσης. για να μπορέσουμε να ακούσουμε ήσυχα τον Επίτροπο τον υποψήφιο και πρώτα Καλώς ορίσατε όλοι στη δημόσια αυτή ακρόαση. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας θέλω να ε, καλωσορίσω τον κύριο Μίμητσα ε, που έχει προταθεί ως Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο προετοιμάζει ε, την εκλογή της Νέας Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 118 και το παράρτημα 16 του κανονισμού μας. Ε, αξιολογώντας όλους τους τα επιτρόπους βάσει της γενικών ε, προσόντων, την ευρωπαϊκή προσήλωση και προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης, εκτιμά το Κοινοβούλιο και αξιολογεί την κατανόησή του και τη γνώση του για το χαρτοφυλάκιο, καθώς επίσης και τι επικοινωνιακές τους ε, δεξιότητες. Η παρούσα ακρόση έχει αυτό το σκοπό, είναι δημόσια και μεταδίδεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και από το Europe by Satellite. Επίσης θα μαγνητοσκοπηθεί η ακρόαση και προσεχώς πολύ σύντομα θα είναι στη διάθεσή σας. Έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες. Έχουμε πολύ αυστηρό χρόνο, αλλά σας παρακαλώ να μιλάτε με κανονική ταχύτητα. Μην προσπαθείτε να μιλήσετε πολύ γρήγορα, υπερβολικά γρήγορα, αλλιώ δεν θα σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Και παρακαλείστε να κλείνετε το μικρόφωνο σας όταν τελειώνετε. Ο προτινόμενος επίτροπος έλαβε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο έχει απαντήσει γραπτός, έχετε λάβει όλοι τις γραπτές απαντήσεις και διατίθενται επίσης ε, και στην Θα σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία. Πρώτα, ο, ο προτινόμενος επίτροπος θα κάνει την εισαγωγική του δήλωση που δεν θα υπερβεί τα 15 λεπτά. Η βασική ε, ακρόαση συνίσταται σε 45 ερωτήσεις από τους βουλευτές. Στο πρώτο γύρο θα ακούσουμε ένα εκπρόσωπο από κάθε μία από τις πολιτικές ομάδες οι ερωτήσεις αυτές θα είναι ενός λεπτού, όχι παραπάνω και ο οριστής επίτροπος θα έχει 1,5 λεπτό για να απαντήσει. Μετά από κάθε ερώτηση μπορεί ο ερωτών να κάνει μια σύντομη συμπληρωματική μόνο για 30 δευτερόλεπτα και ο, ο, Οριστή Επίτροπο έχει ένα λεπτό για να απαντήσει. Όλε οι υπόλοιπε ερωτήσει θα είναι του ενό λεπτού και δύο λεπτά η απάντηση. Παρακαλώ να τηρήσουμε πάρα πολύ αυστηρά το χρόνο μα, διότι δεν έχουμε ε, πολύ χρόνο. Θα έχουμε και δύο ερωτήσει από άλλε προσκληθήσει επιτροπέ, που είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή ε, Διεθνού Εμπορίου. Μετά τους συντονιστές θα λάβουν το λόγο και μετά ε, θα ακολουθήσουν οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Αυτά είναι τα διαδικαστικά. Ελπίζω να πάει καλά η ακρόαση και με την ησυχία μας και ήσυχα να αφήσουμε τον κύριο Μίμητσα να μιλήσει. Έχετε το λόγο παρακαλώ για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έρχομαι στην Επιτροπή σα ω προτινόμενο Επίτροπο για το φυλάκιο τη Διεθνού Συνεργασία και τη Ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εξωτερική δράση. Πρωταρχικό τη στόχο είναι να μειώσει και μακροπρόθεσμα να εξαλείψει την φτώχεια. Είναι μια πολιτική για τον κόσμο, για του πολίτε και ενισχύει την αλληλεγγύη, στηρίζεται σε αυτή γιατί είναι πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών αλληλεγγύη με του ανθρώπου που ζουν με λιγότερο από ένα ευρώ τη μέρα και ρισκάρουν τη ζωή του για να φτάσουν σε ευρωπαϊκέ ακτέ με σχεδίες που και σαπιοκάραβα που συχνά γινόνται και τα φέρετρά του. Αλληλεγγύη προ τι γυναίκε, που είναι θύματα σεξουαλική βία ή ανθρώπου που διώκονται επειδή ανήκουν σε μειονότητε. Ε, αλληλεγγύη προς τα παιδιά στρατιώτε. Η αναπτυξιακή πολιτική αποσκοπεί στην εταιρική σχέση που στηρίζεται σε αμοιβέ συμφέροντα. Όταν ευάλωτα κράτη καταραίουν ή εξαπλώνεται η τρομοκρατία στην Αφρική, αυτό δημιουργεί άμεση απειλή για την Ευρώπη. Όταν αυξάνονται οι εμπορικέ ροέ και βελτιώνεται το κλίμα για τι επιχειρήσει, δημιουργούνται ευκαιρίε και για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταπληκτικέ επιδόσει στην αναπτυξιακή πολιτική. Μαζί με τα κράτη-μέλη αποτελεί το μεγαλύτερο δωρητή παγκοσμίω, προσφέροντα ένα του ίμιση του συνόλου τη αναπτυξιακή βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο των αναπτυσσομένων χωρών, καθώ και βασική πηγή τεχνολογία, καινοτομία, επενδύσεων και επιχειρηματικότητα. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα τη ε, ενίσχυση και στην συνεκτικότητα τη αναπτυξιακή πολιτική. Αν, αν με εγκρίνετε ω Επίτροπο, δεσμεύομαι να αφιερώσω την εμπειρία μου και να, να προσιλωθώ προκειμένου να εξασφαλίσω τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή, αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα έχει κέρια, ε, σημασία για το πρόγραμμα μετά το 2015 και τις διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο μετά τη διαδικασία Κοτονού και φυσικά για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής. Φτάνουμε στην πρώτη προτεραιότητα, ένα φιλόδοξο πλαίσιο μετά το 2015. Οι ισχύοντες αναπτυξιακές στόχοι της χιλιετίας ε, απέφεραν ε, εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενθαρρυντικά για τη μείωση της ε, φτώχεια που έχει μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στο μισό. Σήμερα πολύ λιγότεροι άνθρωποι πηγαίνουν να κοιμηθούν νηστικοί, λιγότερα παιδιά πεθαίνουν από αρρώσεις που μπορούμε να προλάβουμε και όλο και περισσότερα παιδιά, ιδιαίτερα κορίτσια, ε, παρακολουθούν ε, σπουδές. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στι δάφνε μα. Μία γυναίκα στην Αφρική έχει 29, 29 ε, περισσότερες 29 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Περίπου 750 εκατομμύρια στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλέ πόσιμο είδωρ. Και δυστυχώ ε, η φτώχεια είναι ακόμη μια συγκλονιστική πραγματικότητα. Πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο πεθαίνουν από υποσυτισμό και λιμοκτονούν. Φυσικά υπάρχουν και αυξανόμενες ανισότητες και γεωγραφικά χάσματα. Και ενώ η Ασία και η Λατινική Αμερική βρίσκονται σε πιο καλό δρόμο, η υποσαχάρης Αφρική υστερεί. Πάνω από 120 εκατομμύρια διαβίουν σε απόλυτη φτώχεια, περισσότεροι από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Το πλαίσιο μετά το 2015 θα πρέπει να συμβάλλει στην εξάλληψη της φτώχειας και να συμβάλλει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να σταματούμε τη φτώχεια στη ρίζα της, το κακό στη ρίζα του. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση και να βρει την βέλτιστη ισορροπία μεταξύ τους. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου, καθώς και της ειρήνης και της ασφάλειας. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση να συνδυάσουμε όλες αυτές τις πτυχές και να τις εντάξουμε σε ένα ενιαίο, οικουμενικό και περιεκτικό πλαίσιο που θα ισχύει για όλες τις χώρες τις πλούσιες και τις φτωχές. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ε, υλοποιήσουμε αυτή την πρόκληση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να διαμορφώσουν κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και να αναλάβουν την ευθύνη το, της ανάπτυξής τους. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για κάποιον άλλον είναι όχι να μοιραστούμε τα πλούτη μας, αλλά να του δείξουμε ποιος είναι ο δικός του πλούτος. Βασικό στοιχείο της διαδικασίας μετά το 2015 θα είναι η ανάπτυξη της χρηματοδότησης και κυρίως των μέσων εφαρμογής. Συμφωνώ πλήρως με τον, πρόεδρο, τον πρόεδρο Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε στις, στους στόχους της χιλιετίας και να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να, να, επενδύσουν τουλάχιστον 0,7% του ΑΕΠ τους στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό το στόχο και να τον υλοποιήσουμε μέχρι το 2015, κάτι που προς το παρόν είναι ανέφικτο. Αναγνωρίζουμε βέβαια τα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων χωρών της Ευρώπης, αλλά θα ήθελα να απευθύνω έκλειστα στα στο νέο πλαίσιο να τηρήσουν αυτή την υπόσχεση. Για να βελτιστοποιήσουμε την επίπτωση της ενίσχυσης θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά της επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο συντονισμό και στην καλύτερο, καλύτερο συνδυασμό της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να αυξήσουν τους εθνικούς τους πόρους με χρηστή οικονομική διαχείριση, καλύτερη διακυβέρνηση, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και με αποτελεσματικά και δίκαια φορολογικά συστήματα. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιήσουν κάποια καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στην αξιοπρεπή εργασία. Μόνο με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, όπου όλοι οι συμβαλόμενοι θα παίζουν τον ρόλο τους, θα οδηγηθούμε στην επιτυχία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, προκειμένου να υιοθετήσει μια, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη συνολική ελληνική και την εξασφάλιση ενός αηφόρου μέλλοντος που δεν θα αποκλεί κανέναν. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να εγκαινιάσω και να διαπραγματευτώ ένα πλαίσιο για μετά τη Συμφωνία Κοτονού και μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Αφρική. Η υφιστάμενη Συμφωνία Κοτονού είναι η πιο περιεκτική συμφωνία βορρά-νότου στον κόσμο. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση. Βέβαια, οι χώρες εκεί είναι πολύ σημαντικές για μας περισσότερο από ποτέ θα έλεγα. Το θέμα είναι πώς θα διαμορφώσουμε και θα σχεδιάσουμε καλύτερα τη συνεργασία μας στο μέλλον. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να αντικατοπτρίζει την έκβαση της διαδικασίας μετά το 2015. Δεν μπορεί να αποτελεί μια απλή συνέχιση του παρελθόντος. Η ομάδα των χωρών ΑΚΕ επίσης σκέφτεται την ε, συνέχεια της διαδικασίας και εμείς θα πρέπει το, να κάνουμε το ίδιο ενισχύοντας την εταιρική μας σχέση με τις χώρες ΑΚΕ φυσικά με βάση το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε ε, των χωρών και των περιφερειών. Θα πρέπει από κοινού να συζητήσουμε πώ θα προωθήσουμε την εταιρική μα σχέση. Ω πρώτο βήμα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια ευρεία διαβούλευση και διάλογο τα επόμενα χρόνια. Η τρίτη μου προτεραιότητα είναι να συμβάλλω σε μια μεγαλύτερη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Γιατί ο κόσμος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ε, της ειρήνης, της ασφάλειας, της ενέργειας, των κλιματικών αλλαγών, της γεωργίας και του εμπορίου. Μεγαλύτερη συνοχή λοιπόν των εσωτερικών και εξωτερικών μας πολιτικών αποτελεί επιτακτική ανάγκη εκ των όνων προϋπόθεση και η συνεργασία που θα προσφέρουμε στους εταίρους μας δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια αμυγή βοήθεια, αλλά να περιλαμβάνει θέματα όπως επιστήμη, υγεία, εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, νεολαία, εργασιακή κινητικότητα και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι θα πρέπει να περιλάβουμε νέα στοιχεία στο σχεδιασμό των πολιτικών μας. Ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ε, συνοχή των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η δομή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συμφωνία στη, μεθοδολογία εργασίας με την ΥΠΑΤΗΚ εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο, καθώς και τους υπόλοιπους επιτρόπους, θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνεργειών και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών μας. Προσωπικά θα συμβάλλω στην υλοποίηση αυτών των προσπαθειών. Η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, την, την πολιτική ανθρωπιστική βοήθεια, την εμπορική, την μεταναστευτική και άλλε πολιτικέ. Αν εγκρίνεται ε, την. Αν με εγκρίνεται ως επίτροπο θα προσπαθήσω να συμβάλλω στην συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και να έχω στενή συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Επίσης, ε, θα παρακολουθώ την υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών και θα έχουμε συνεργασία σε πρώιμο επίπεδο με τους υπόλοιπους επιτρόπους προκειμένου να προβούμε σε μία ενδελεχή ανάλυση των πρωτοβουλειών μας. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι ε, Ευρωβουλευτή κυρία Πρόεδρε, 83% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους, τις αναπτυσσόμενες χώρες. 61% των συμπολιτών μας πιστεύουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια και 70% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η προσφορά ρογής σε αναπτυξόμενες χώρες έχει και για αυτούς θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής και να προβάλλουμε περισσότερο τα επιτεύγματά μας. Γι' αυτό και θα ήθελα μία πολιτική που να είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα και να πιάνει τόπο το κάθε ευρώ. Το επόμενο έτος θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Θα είναι ιδανική ευκαιρία να έχουμε επαφή και διάλογο με τους πολίτες και να εξηγήσουμε πώς η αναπτυξιακή μας πολιτική είναι επωφελής για όλους μας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, αν επιβεβαιώσετε την, το διορισμό μου, θα συνεχίσω να επιδιώκω στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά θα τιμήσω τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο στρατηγικό και διορθωμένο διάλογο και θα επιδιώκω τακτικό και τακτικό άτυπο διάλογο μεταξύ μας. Τέτοιος διάλογος θα είναι πολύ σημαντικός ε, για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε ε, θετικά την διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού πλαισίου μετά το 2015 και να ε, αποφαινόμαστε με ενιαφωνή και να προασπίζουμε ένα ενιαίο όραμα. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Μίμητσα. And for sticking very well to your time. Ε, τηρήσατε και θαυμάσια το χρόνο σας και σας ευγνωμονώ γι' αυτό. Αρχίζουν οι ερωτήσεις τώρα. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Στήρα από το ΕΛΚ πρώτος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μιμίτσα, και εσείς ο ίδιος είπατε ότι εφόσον επιβεβαιωθεί ο διορισμός σας, από τα σημαντικότερα θέματα που θα σας απασχολήσουν είναι οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο μετά το 2015. Και μάλιστα η ομάδα εργασίας ήδη προ... πρότεινε ένα σχέδιο για τους επόμενους μελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας Βέβαια, αν έχουμε πολλέ προτεραιότητε, είναι σαν να μην έχουμε καθόλου προτεραιότητε. Αν μπορείτε να επικεντρωθείτε σε λίγε από αυτέ, σε ποιε προτεραιότητε θα δίνατε ε, έμφαση. Ωραία. Μου δίνετε και μία μεγάλη ευκαιρία και να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα κροατικά. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την ευκαιρία και ε, θα την έχουμε πολύ πιο συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη φάση λοιπόν της προετοιμασίας του σχεδίου για, την, για τους επόμενους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, ε, θα ήθελα να πω ότι τα κράτη-μέλη συνέβαλαν τα μάλα στη διαδικασία αυτή. Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο για τους μελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους που θα αποτελέσει τη βάση για την συνέχεια των εργασιών. Τώρα, η προσωπική μου θέση είναι ότι σε ό,τι αφορά τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης, Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στον περιορισμό των προτεραιοτήτων, ώστε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους στόχους. Γιατί πραγματικά αν έχουμε ε, μια πληθώρα στόχων θα έχουμε πολλές αποσπασμένες προσπάθειες και έτσι δεν θα επικεντρωθούμε στην αηφόρο ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε πολύ περιορισμένο αριθμό στόχων. Και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση, δηλαδή να περιορίσουμε τους στόχους μας σε μικρό αριθμό προτεραιοτήτων και σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, σε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Και αυτοί οι λίγοι περιορισμένοι στόχοι να προσδιορίσουν το περιεχόμενο της μελλοντικής μας εργασίας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Σίγουρα είναι πολύ ε, δύσκολο αυτό το έργο, γιατί το να προσδιορίσετε συγκεκριμένου στόχου και να περιοριστείτε σε συγκεκριμένου στόχου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσετε άλλου, αυτό απαιτεί τη λήψη τη, πολύ σοβαρών αποφάσεων. Μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι στη διαδικασία αυτή θα έχετε στενή συνεργασία και διαβουλεύσεις με τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Ανάπτυξη και γενικώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μια άλλη ερώτηση με ποιο τρόπο στην διαπραγματευτική στρατηγική θα αναζητήσουμε εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να καταφέρουμε επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτό που έχουμε ενώπιό μας και στο οποίο θα φωσιωθώ πλήρως εφόσον εγκριθεί η υποψηφιότητά μου είναι να επικεντρωθούμε σε σαφείς στόχους που θα γίνουν δεκτοί από, όλες, από όλους τους ε, συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε δηλαδή στόχους ε, που κυρίως επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, γιατί ο στόχος αυτός ακόμη δεν βρίσκεται στο επίπεδο των φιλοδοξιών των ε, χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό το στόχο. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα κατάλληλα μέσα για την ε, υλοποίηση όλων των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα διασφαλίσουν, και θα φροντίσω και εγώ γι' αυτό, θα διασφαλίσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο, και, ώστε και οι δύο στόχοι να προσδιοριστούν με όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένο τρόπο γίνεται και με συγκεκριμένες δράσεις. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία τις σχετικές εκθέσεις για την ανάπτυξη των μελλοντικών μας στόχων από την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ κύριε Μίμητσα από τους σοσιαλιστές. Τώρα, ο κύριος Λίτς. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δήλωσή σας και την εισήγησή σας. Η τρέχουσα κρίση του έμπολα στην Δυτική Αφρική δείχνει ότι η απάντηση ήρθε πολύ αργά και ότι έλειπε ο κατάλληλος συντονισμός. Τα υγειονομικά συστήματα δεν έχουν τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν επιδημίες. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εισήγαγε ένα, μια ανακοίνωση για ένα νέο ρόλο στην παγκόσμια υγεία που ενισχύει την ε, καθολική υγειονομική περίθαλψη. Εσείς θα συνεχίσετε αυτή την εργασία και θα προτείνετε κάποιο πρόγραμμα για δράση, ιδιαίτερα για τις χώρες νοτίως της Σαχάρα που υποφέρουν ε, περισσότερο από τις επιδημίες από ότι όλα τα υπόλοιπα κράτη στον, κόσμο. Αυτό σημαίνει ε, απάντηση, ταχύτερη δηλαδή ανταπόκριση σε περιπτώσεις ξεσπάσματος επιδημίας όπως η τωρινή του έμπολα και συμφωνείτε πως σαφής ε, ηγετική ικανότητα αλλά και συντονισμός των δωρητών είναι απαραίτητο ε, για να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Για το έμπολα και την ε, κρίση του έμπολα, την επιδημία του έμπολα, θα έλεγα ότι το επίγον είναι να απομονωθεί η αρρώστια και όχι οι χώρες όπου έχει εκδηλωθεί η επιδημία. Ε, η απάντησή μας αυτή τη στιγμή σχετίζεται περισσότερο με την ανθρωπιστική πτυχή της ευρωπαϊκής δράσης εξορισμού ε, συμβαίνει αυτό, διότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αυτή που χρειάζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ε, ταυτόχρονα όμως το έμπολα αποτελεί την ευκαιρία και την πρόκληση για να σκεφτούμε μια συνεπή σύνδεση ανάμεσα στην αποκατάσταση, την ανακούφιση και τις αναπτυξιακές πολιτικές με συνεπή τρόπο. Θα έλεγα ότι αυτή η εμπειρία θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη στο να δημιουργήσει ε, συντονισμό και συνοχή. Συμμετέχουμε οικονομικά με πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ βοηθώντας ε, την ε, αντοχή των υγειονομικών συστημάτων των χωρών που πλήττονται από την επιδημία αλλά ε, πρέπει να ε, δοθεί και μη οικονομική βοήθεια ε, με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και γιατρών επιτόπου αλλά και συντονισμός με τους άλλους δωρητές και άλλους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ ο κύριος Λίτζ. Η επόμενη ερώτηση μάλλον είναι η εξή. Τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όπως, ε, μάλλον περιλαμβάνουν μεγάλα προβλήματα όπως το AIDS, η θνησιμότητα ε, των μητέρων. Τα δικαιώματα όμως αυτά ε, πλήττονται περισσότερο στις ευάλωτες μερίδες των πληθυσμών. Εσείς συμφωνείτε ότι θα έπρεπε αυτά τα δικαιώματα να συμπεριλαμβάνονται στην καθολική υγειονομική περίθαλψη και στις κυβερνητικές πολιτικές και ότι η Ένωση θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο ώστε να δώσει τα δικαιώματα αυτά στις ε, κοινωνίες που πλήττονται. Μάλιστα. στο πρόγραμμά μας για τις δραστηριότητε μας και για τις απαντήσεις μας στις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη Διαρκώς τονίζουμε ότι ο τομέας της υγείας είναι ένας πολύ σημαντικός ε, τομέας αυτής της βοήθειας. Η οικοδόμηση ενός υγειονομικού συστήματος, το οποίο θα είναι για όλους, αλλά και θα προσφέρει υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρο τον πληθυσμό κάθε αναπτυσσόμενης χώρας είναι ο τελικός μας στόχος, ο απότερος μας στόχος. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν καλούμε στο πρόγραμμα δράσης που ακολουθεί τη διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ε, ε, δημογραφική κατάσταση στο Κάιρο είχε γίνει Καλούμε λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες να τοποθετήσουν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τα σεξουαλικά δικαιώματα ε, στο, στην πρώτη προτεραιότητα. Και αυτό θα είναι το πρώτο τμήμα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Βοήθειας και Ανταπόκρισης. Σας ευχαριστούμε κύριε Λίτς και κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε. Και τώρα ο κύριος Λούκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε, θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ γενική ερώτηση για το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τον εαυτό σας στη νέα σας θέση. Η αναπτυξιακή πολιτική είναι κάτι που γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Και υπάρχει και ευρωπαϊκή Σύμφωνα όμως με την αρχή της επικορικότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλύπτει μόνο εκείνους τους τομείς και να προωθεί που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο παρά μόνο σε ευρωπαϊκό. Οπότε, θα σας παρακαλούσα συγκεκριμένα να μας πείτε σε ποιους τομείς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει καλύτερα και να ασκήσει καλύτερα αναπτυξιακή πολιτική από ό,τι μπορούν τα κράτη-μέλη. Παρακαλώ συγκεκριμένα να μας αναφέρετε κάποιους τομείς και μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει με την απάντηση που δώσατε στην πρώτη ερώτηση προηγουμένως. Είπατε ότι θέλετε να περιορίσετε τον αριθμό των στόχων και να ε, τους κάνετε πιο συγκεκριμένους για την αναπτυξιακή πολιτική. Ποιοι είναι δηλαδή εκείνοι που θα εγκαταλείψετε τελείως ή δεν θα τους ε, Δώστε τόση μεγάλη ε, προσοχή. Θα τους αναθέσετε στην επικουρκότητα στα κράτη-μέλη και θα επικεντρωθείτε στους στόχους που μπορείτε να αποδείξετε ότι είναι καλύτερα σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα διεκπεραιώνει αυτά από ότι τα κράτη μόνα τους. Και ποιοι είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι στόχοι. Ε, for me, development policies... Για μένα η αναπτυξιακή πολιτική και ιδιαίτερα η αηφόρος αναπτυξιακή πολιτική νοείται ως μια πολιτική που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα δικαιώματα ε, και στα συμφέροντα της επικουρικότητας των κρατών μελών. Μιλούμε για συνοχή πάντα της αναπτυξιακής μας πολιτικής και δεν εννοούμε μόνο ε, τις εσωτερικές πολιτικές στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη αλλά εννοούμε και το συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων ε, κρατών και των διαφόρων δωρητών και χορηγών. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο το βλέπουμε ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τον επικείμενο γύρο ε, για τον συντονισμό της αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει ακριβώς να είμαστε πολύ στοχευμένοι στη δράση μας για να αντιμετωπίσουμε τους στόχους της ανάπτυξης. Και το πλαίσιο που έχει οριστεί για τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι η επικουρικότητα είναι κάτι το οποίο είναι αποσπασμένο από την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική. Υπάρχει και χώρος και πολλοί λόγοι να συνεργαζόμαστε, να συντονίζουμε τις δραστηριότητες των οριτών και με τρόπο που θα αντανακλά και τα συμφέροντα και των κρατών μελών και τις ίδιες τους τις δράσεις. Είναι συμπληρωματικές αυτές οι προσπάθειες. Συμπληρωματική επερώτηση έχετε, κύριο Λούκε. Ναι. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Ich hatte Σας παρακάλεσα συγκεκριμένα να μας δώσετε στόχους. Τώρα μιλήσατε για συνεργασία, για συντονισμό, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια φωνή. Δεν είναι συγκεκριμένα όλα αυτά. Σας παρακάλεσα να μας δώσετε συγκεκριμένους στόχους της ε, ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής που βλέπετε συγκριτικό πλεονέκτημα από το γεγονός ότι ασκεί ε, αυτή την πολιτική και βάζει αυτούς τους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν γίνεται καλύτερα ε, σε επίπεδο κρατών μελών. Άγω... Θα ε, ήθελα να σας αναφέρω ορισμένες δράσεις και τομείς, ε, έτσι, να τονίσω για την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική και πιο ε, στοχευμένη σε αποτελέσματα από τις μεμονωμένες προσπάθειες και συνεισφορές των κρατών μελών. Παράδειγμα, όταν μιλούμε για χρηστή διακυβέρνηση, και όλο τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αιρεσιμότητα, δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις που βάζουμε ε, για χρηματοοικονομική υποστήριξη και προγράμματα τέτοια. Μπορούμε ως Ευρώπη να έχουμε καλύτερες επιδόσεις από τα κράτη-μέλη ξεχωριστά. Στον πολιτικό διάλογο έχουμε δυνατότητα μεγαλύτερης επιρροής για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στι αναπτυσσόμενες χώρες καλύτερα και σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από ό,τι θα έκαναν μεμονωμένα τα κράτη-μέλη. Ακόμα και στον τομέα της υγείας ή της παιδείας. Μια κοινή ευρωπαϊκή δράση, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, θα ήταν πιο αποτελεσματική από ότι η μεμονωμένη και ίσως αποσμασματική δράση των κρατών μελών. Ευχαριστώ από τους φιλελευθέρους ο κύριος Γκέρενς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αφήξω ένα θέμα σε σχέση με την ε, χρηματοδότηση της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Το θέμα είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που έχουν καταστεί απαραίτητα ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών. Την περασμένη εβδομάδα, ένα εκπρόσωπο τη Κομισιόν δήλωσε ενώπιον τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή ότι τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό τη ανάπτυξη. Το να μην γίνει κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ναρκοθέτηση τη καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όμω είμαστε τη άποψη εδώ και χρόνια σε αυτή την επιτροπή ότι το να δοθούν τα χρήματα ε, κατά μάλλον το να βαρύνουν τα χρήματα των κλιματικών αλλαγών τον αναπτυξιακό προπολογισμό ε, ε, ε, τροχοπεδούν την καταπολέμηση της στόχιας. Ποια είναι η δική σας άποψη και ε, τι θα κάνετε για να επηρεάσετε την, επηρεάσετε την υπόλοιπη Επιτροπή πριν ληφθεί απόφαση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η συζήτηση για την αύξηση των κονδυλίων που στόχο έχουν την αντιμετωπίση των κλιματικών αλλαγών ίσως να έχει έρθει κάπως αργά, διότι το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει ήδη, έχει εγκριθεί από όλους τους αρμόδιους σε αυτή τη διαδικασία και αυτό που έχουμε ενώπιόν μας είναι μια ε, κοινή κλιματική, ε, μια διάσκεψη μάλλον για τις κλιματικές αλλαγές όπου θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια οικονομική δέσμευση. Τώρα όμως ε, εξετάζοντας το χαρτοφυλάκιο της ανάπτυξης βλέπω πως το 20% της αναπτυξιακής βοήθειας του κονδυλίου του αναπτυξιακού ας το πούμε έτσι ήδη κατευθύνεται ε, ε, ε, στις, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό είναι εντό, είναι εφικτό και ίσως να μπορέσουμε να δώσουμε και κάπως περισσότερο από ότι 20% από το μέσο το αναπτυξιακό, το EDF. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε πώς οι κλιματικές αλλαγές ε, θα σχετιστούν και με άλλα κομμάτια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πάντως θα πρέπει να βρούμε μη παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό που έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι όταν φτάσουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς, θα πρέπει σαφώς να λάβουμε υπόψη την χρηματοδότηση για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και βεβαίως θα έχω διάλογο και με το Κοινοβούλιο και με τη δική σας Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ που δείχνεται διαθεσιμότητα ε, να συζητήσετε με την Επιτροπή μας για αυτά τα θέματα είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσετε και πολύ θα το θέλαμε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να αποφευθεί είναι να παρακολουθήσουμε την, μια παράλογη κατάσταση όπου θα έπρεπε να ξαναδοθούν πόροι ε, που έχουν δοθεί ε, με στόχο την καταπολέμηση της στόχης να δοθούν αλλού, να πρέπει να τοποθετηθούν αλλού, δηλαδή στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Γι' αυτό σας έθεσα αυτή την ερώτηση και ξεπανερχόμενο στη διαθεσιμότητά σας ήθελα να δω σε ποιο πνεύμα αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα και αν είστε έτοιμος να προσεγγίσετε περισσότερο την άποψη της δικής μας εδώ Επιτροπής. Ναι, μάλιστα. Ε, δυστυχώς ε, οι πιστώσεις πληρωμών και υποχρεώσεων αλλά και οι περιορισμοί που τις περικλείουν μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσε κανείς να δει πως υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στους αναπτυξιακούς στόχους και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όμως, σε ένα βιώσιμο πλαίσιο δεν θα πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση, διότι είναι κοινός, ε, ε, κοινή η δράση που χρειάζεται. Οι κλιματικές αλλαγές είναι σημαντικές και αποτελούν τμήμα του βιώσιμου πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα βρίσκομαι σε συζήτηση με το Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση εντός των ορίων που δυστυχώς μας επιβάλλονται λόγω του πολιτούς προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάντσες Καλδεντέη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Η πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη είναι μια γενική αρχή που θα πρέπει να διέπει όλες τις πολιτικές ένωσες που έχουν επίδραση στις αναπτυσσόμενες χώρες και στους λαούς τους. Και αν ε, δεν ε, ενισχύσουμε τέτοιες πολιτικές, ε, θα έχουμε πολλούς κερδισμένους και πολλούς χαμένους και αύξηση των ανισοτήτων. Θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη, να εξασφαλίσουν τη συνοχή των πολιτικών, των αναπτυξιακών πολιτικών, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος πριν από λίγο. Η ερώτησή μου είναι εξής. Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να πρωτοστατήσει σε μια διαδικασία διατησίας και να είναι αρμόδιος ώστε να κρίνει κατά πόσο υπάρχει συνοχή μεταξύ των πολιτικών που ανήκουν στα χαρτοφυλάκια διαφόρων επιτρόπων. Φυσικά πρέπει να έχουμε συνοχή μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των πολιτικών που εμπίπτουν στους τρεις πυλώνες ε, της αηφόρου ανάπτυξης, ε, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Και η ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων είναι πολύ σημαντική. Δεν θα πρέπει να αδιαφορήσουμε για κανένα από αυτούς τους τομείς. Δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε κανένα τομέα. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε το στόχο μας στην καταπολέμηση και μακροπρόθεσμα την εξάλληψη της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα μπορούσαμε και θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια μόνο εφόσον υιοθετήσουμε μια συνεκτική προσέγγιση μεταξύ των τριών πυλώνων που ανέφερα. Γιατί η, μόνο η οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να αυξήσει όπως φαίνεται, να ενισχύσει τις ανισότητες μεταξύ των χωρών γιατί υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες ανισότητες στην ανάπτυξη και όλο και περισσότερη φτωχή. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και τους άλλους δύο πυλώνες για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανεκτικότητά τους και προσαρμοστικότητά τους. Σίγουρα και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι Αντιπρόεδροι θα πρέπει να συντονίζουν την κατάσταση και φαίνεται και από την παρουσίαση του προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκανε ο πρόεδρος Γιούγκερ. Ζητούμενο είναι μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε όλες οι πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες και την ε, εξασφάλιση της αηφορίας τους. Δεύτερη ερώτηση ακολουθώντας τον ερμό της πρώτης. Τι μηχανισμούς ε, ε, ζήτησης θα δημιουργήσετε ώστε να δώσετε ενάυσματα και στους τοπικούς αλλά και στους εθνικούς φορείς να κάνουν καταγγελίες ή να απευθύνουν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαφάνεια και η ανοιχτή στάση της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, είναι μια εξελικτική διαδικασία που συνεχώς ε, βελτιώνεται. Η διαφάνεια είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Και αυτό ισχύει και για τον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το θέμα στην αναπτυξιακή συνεργασία, γιατί έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ε, σχέδια και προγράμματα στα οποία συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, τοπικοί φορείς, ε, τοπικές αρχές και πολλοί άλλοι παράγοντες. Γι' αυτό και θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή κάθε προγράμματος μεμονωμένου και να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη μηχανισμών ή διαδικασιών ώστε να μην περνάνε παρατήρητε τα προβλήματα και να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής ή υποβολής καταγγελιών για τις διάφορες φάσεις εφαρμογής ενός προγράμματος. Πάντως, το ποσοστό σφάλματος που ισχύει αυτή τη στιγμή, που είναι γύρω στο 2 με 3% δεν είναι και πολύ χαμηλό, Παρ' όλα αυτά, 97% των προγραμμάτων και σχεδίων μας που εφαρμόζονται σε δύσκολες καταστάσεις και σε αδίξιες συνθήκες και σε επικίνδυνα περιβάλλοντα διέπονται από διαφάνεια και καθορίζονται από ε, τους στόχους της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα από τους Πρεσίνους τώρα. Ευχαριστώ πολύ οριστέντα επίτροπε, προφανώς θέλετε να φέρετε και την ιδιωτική οικονομία πιο κοντά στην αναπτυξιακή βοήθεια της επιχειρήσης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, θα υποστηρίζατε δεσμευτικού κανόνες και κοινωνική εταιρική ευθύνη έτσι ώστε στο μέλλον να ακούμε λιγότερα θλιβερά όπως οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην κλωστοϊφαντουργία στο Μπαγκλαντές ή σε άλλους κλάδους που απασχολούν παιδιά και θα ήσασταν πρόθυμος να περάσετε ε, πέρα από ένα σύστημα συμφωνίας κυρίων και μη δεσμευτικών ε, εθελουσίων ε, συμφωνιών και μετά το 2015 πώς σκέφτεστε να εγγράψετε αυτούς τους στόχους στην ε, ατζέντα, την αναπτυξιακή. Ευχαριστώ πολύ. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα ε, καθίσταται όλο και πιο πρωταγωνιστικός για να βελτιωθούν οι δράσεις ε, και στις χώρες εταίρους μας, οι αναπτυξιακές εννοώ, αλλά και στα δικά μας αναπτυξιακά προγράμματα για τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό απαιτεί όλο και περισσότερο αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και όντως αναλαμβάνουμε κάποιες δράσεις ε, και αρκετές για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοινωνική εταιρική ευθύνη με το πιο διαφανή και σωστό τρόπο. Παράδειγμα, έχουμε μια πρωτοβουλία αυτό τον καιρό για ε, ε, εξόριξη ε, διαμαντιών ή μεταλλευμάτων σε χώρες που βρίσκονται στη σύραξη και κάποια αντίστοιχα θέματα Πολύ σύντομα θα επαναξετάσουμε την κατάσταση που ισχύει για να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε αντιμέτωποι με τις ευθύνες της και την κλωστοεφαντουργία ε, σε περίπτωση που είναι χαμηλές οι προδιαγραφές, ε, τα πρότυπα εργασιακά ή ε, η απασχόληση παιδιών. Είναι πιο συγκεκριμένα και ειδικά θέματα αυτά. Θα συζητήσουμε ευθέτω χρόνο με την Επιτροπή σας παραδέχομαι ότι παραμένει όντως εθελοντική αυτή η δράση και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Να αφήσουμε ε, κάποια χρονική περίοδο για να αποτιμήσουμε από κοινού τα αποτελέσματα αυτής της εθελοντικής προσέγγισης και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε πιο δεσμευτικές ρυθμίσεις, νομικά δεσμευτικές για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Uh, ε, ερώτηση. Γνωρίζω ότι έχετε, ε, προέρχεστε από το εμπόριο και έχετε εμπειρία σε αυτό το κλάδο, πράγμα πολύ χρήσιμο. Τι ε, θα κάνετε με τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες για να αποφύγουμε τόσο θλιβερά και δυστική, ε, ατυχή ε, φαινόμενα όπως είναι η παραβίαση δικαιωμάτων αυτοχθών λαών, η αρπαγή της γης τους ε, και άλλοι παραδοσιακοί χρήστες γης βλέπουν τη γη να φεύγει από τα χέρια τους όταν έρχονται μεγάλοι επενδυτές να εγκατασταθούν στη χώρα. Πώς θα δείξετε έτσι περισσότερο οξύ αντίδραση. Η αναπτυξιακή πολιτική και τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι ήδη αλλά και στο μέλλον θα είναι ακόμα περισσότερο προσανατολισμένα στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Θέλουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις χωρίς αποκλεισμούς όμως, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να, να δραστηριοποιούνται και οι μικρομεσαίοι στην αναπτυξιακή βοήθεια και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεσμεύομαι πραγματικά εδώ να εμβαθύνω σε αυτή την προσπάθεια και σε προγράμματα που θα βοηθούν για την καλύτερη διακυβέρνηση και να επιτρέπουν να γίνονται σεβαστά τα δικαίωματα ιδιοκτησίας γης για τους μικρούς ε, κτηματίες, πούμε, όχι τους μεγάλους, τις μεγάλες εταιρείες που αρπάζουν τη γη από τους αυτόχθονες. Ας αρχίσουμε λοιπόν εκεί από τη συμπεριλήψη της άτυπης ακόμα ε, οικονομίας, ιδιαίτερα στη γεωργία σε αυτή την προσπάθεια. Να μην βοηθούμε και να διευκολύνουμε τη δράση των μεγάλων εταιρείων που έχουν έτσι επιθετική επενδυτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράο από το EFTD. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το διεθνές εμπόριο είναι ένας από τους τομείς όπου η λέξη συνοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι πολυμερείς και οι διμερείς συμφωνίες πολύ συχνά επηρεάζουν βία την κοινωνικό ιστό και την ανάπτυξη. Μία στενή επαφή με τον Επίτροπο Ανάπτυξης θα πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε το εμπόριο να στηρίζει το βιώσιμο, τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, και να υπάρχει συνοχή. Εγώ ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να συμμετέχετε ε, δραστήρια στις εμπορικές διπλωματεύσεις με τις τρίτες χώρες και σκοπεύετε να συμμετέχετε όντως και να παρέμβετε στην ε, ατζέντα των πολυμερών διαπραγματεύσεων. Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβετε ώστε να εξασφαλίσετε ότι η εμπορική πολιτική εν γέννη θα εγγυώνται τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αναπτυξισόμενες χώρες και δεν θα ε, ε, ε, καθυστερήσουν αντίθετα την ανάπτυξή τους. Ευχαριστώ. Link between development and trade is one of... Η ανάπτυξη και το εμπόριο είναι όντως είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία συνοχής για την αναπτυξιακή πολιτική. Σύμφωνα με το σχέδιο το συντονισμού που έχει αναπτυχθεί και που θα θέσουμε σε εφαρμογή μόλις θα πιάσουμε δουλειά, αυτός ο συντονισμός θα μας διευκολύνει να έχουμε αυτή την πολυμερή προσέγγιση στις εμπορικές διαπραγματεύσει και τα εμπορικά ζητήματα στο πλαίσιο της ανάπτυξης, διότι ο Επίτροπος Εμπορίου και ο Επίτροπος Ανάπτυξης θα είναι τμήμα της ομάδας ε, ε, εξωτερικής δράσης και των επιτρόπων που θα συμμετέχουν εκεί υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου. Ε, ε νομίζω λοιπόν πως από εδώ και στο εξή θα είναι πολύ πιο εύκολο και είμαι απόλυτα δεσμευμένος γι' αυτό, ότι δηλαδή η αναπτυξιακή πτυχή, η αναπτυξιακή οπτική ε, και η ατζέντα η αναπτυξιακή της Δόχα θα πρέπει να εντάσσεται μέσα στην ευρωπαϊκή ε, εντολή και την ευρωπαϊκή πολιτική ε, ως βασική για την συμβολή μας στην ολοκλήρωση αυτών των στόχων. Για παράδειγμα, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης που είναι ακόμα υποδιαπραγμάτευση, επίσης θα πρέπει να είναι συνεπής ε, με τους ε, αναπτυξιακούς στόχους. Μάλιστα να κάνω μια πιο συγκεκριμένη και ερώτηση για τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσει του TTIP που είναι η πιο μεγάλη ε, διμερής συμφωνία της ιστορίας και αντιπροσωπεύει το 1 τρίτο του εμπορίου. Θα έχει με τεράστιο αντίκτυπο στις ε, γενικές, ε, γενικούς εμπορικούς κανόνες και στην οικονομία, ιδιαίτερα για τις αναπτυξιακές χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Πώς θα παρέμβετε σε αυτό το πλαίσιο ώστε το εμπόριο να μην θεωρείται πλέον ως ένα όπλο αλλά ως ένα μέσο αναπτυξιακό. Yes, Κατά βάση οι διαπραγματεύσει ανάμεσα σε δύο υπεργούς εταίρους, ε, ναι, τους μεγαλύτερους στον κόσμο όντως, και θα έχει αυτή η συμφωνία τεράστιο αντίκτυπο στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις ε, ανάμεσα στις δύο διαπραγματευόμενες πλευρές. Όμως ε, ο αντίκτυπος αυτός ίσως να επηρεάσει και τις αναπτυσσόμενες χώρες, όχι ποιησίμως δηλαδή ρητός, γιατί είναι διμερείς οι συμφωνίες, ε, σε ισχύωση και περιορίζουν μόνο τα συμβαλόμενα τους μέρη, όμως ε, ως Επίτροπος ε, υπεύθυνο για την Ανάπτυξη ε, δεσμεύομαι να είμαι τμήμα της διαπραγματευτικής ομάδας που πάντοτε θα παρακολουθεί τι αντίκτυπο θα μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε πτυχή της TTIP στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα συμφέροντά τους. Ε, βλέπω τον εαυτό μου ως ένα είδος θεματοφύλακα έτσι ώστε ε, να μην ε, μεταφραστούν, να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις από την TTIP και να μην επηρεάσουν την αναπτυξιακή συνεργασία και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοράου. Έτσι ολοκληρώνει το πρώτος γύρος όπου είχαμε έναν ομιλητή εν ομάδα και τώρα περνάμε στο δεύτερο τμήμα που θα έχουμε τρία λεπτά. Έχουμε δηλαδή ε, μονόλεπτη ερώτηση, δίλεπτη απάντηση και χωρίς επερώτηση πρώτοι δύο ομιλητές προέρχονται από τις επιτροπές που έχουν προσκληθεί σήμερα εδώ. Ο πρώτος είναι από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και είναι ο κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλωσορίζω και τον ε, κύριο Μίμιτσα. Μετά από 1,5 χρόνο έχουμε δεύτερη δυνατότητα ακρόασης και πιστεύω ότι το χαρτοφυλάκιο που σας ανέθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιούνκερ της Αναπτυξιακής ε, Συνεργασίας και Ανάπτυξης πολύ περισσότερο ανταποκρίνεται στην προηγούμενη σας επαγγελματική σταδιοδρομία. Είναι ενδιαφέρον γιατί στη διάρκεια των, της προεκλογικής εκστρατείας ήμασταν ε, σε διαφορετικές πλευρές, αλλά τώρα εσείς εργάζεστε για το δικό μας ε, επικεφαλής υποψήφιο, τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. αυτή είναι και η ομορφιά της ευρωπαϊκής πολιτικής στο, στην επιστολή για την ανάθεση των καθεκόντων σας, ε, ε, ο, ο Επίτροπος Γιούγκερ μίλησε για τις συνεργασίες με την ύπατη εκπρόσωπο Μογκερίνη. Πώς αυτό θα εξασφαλίσει τη συνοχή των ε, πολιτικών τη Ένωση με τις εξωτερικές πτυχέ και τις εξωτερικές πολιτικές και πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσει όπου υπάρχουν ε, κρίσεις όπως η Συρία, το Ιράκ, η έξαρση και η ανάπτυξη της οργάνωσης ίσης και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική ερώτησή σας. Τώρα, η σχέση της εξωτερικής πολιτικής και της ε, πολιτικής ασφάλειας με την αναπτυξιακή πολιτική είναι άρρηκτη. Πρόκειται για αναπόσπαστα συνδεδεμένες πολιτικές και σίγουρα θα πρέπει να αποτρέψουν οποιοδήποτε διαχωρισμό, ιδιαίτερα στις καταστάσεις κρίσης. Και Σίγουρα χωρίς ανάπτυξη δεν έχουμε ασφάλεια και χωρίς ασφάλεια δεν νοείται ανάπτυξη. Στις χώρες που επλήγησαν από εμπόλεμες σειράξεις η φτώχεια είναι 20% ε, μεγαλύτερη από ό,τι σε χώρες που δεν επλήγησαν από τέτοιες ε, συγκρούσεις. Οπότε θα πρέπει να έχουμε συντονισμό και κυρίως του Αρμοδίου Επιτρόπου για την Αναδεξιακή Συνεργασία και της ΥΠΑ της εκπροσώπου ε, της εξωτερικής πολιτικής, που είναι και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό λοιπόν να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο απάντησης, απόκρισης ε, της Ευρώπης σε καταστάσεις κρίσης γιατί πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά εκ των υστέρων σε τέτοιε καταστάσεις κρίση χωρίς να κάνει τον συνδυασμό των διαφόρων στοιχείων και χωρίς να αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό αντίδρασης που έχει. Γι' αυτό ένας ε, συντονισμό ε, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας με την αναπτυξιακή και την ανθρωπιστική πολιτική θα είναι πολύ σημαντικό. γιατί σε πρώτο στάδιο έχουμε εξωτερική πολιτική και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και μετά πιο μακροπρόθεσμα την προσφορά αναπτυξιακής πολιτικής. Ήδη συζητήσαμε το θέμα αυτό του συντονισμού με τον Επίτροπο και συμφωνήσαμε γι' αυτό γιατί υπάρχει τεράστιο δυναμικό τέτοια συνεργασία και συντονισμού. Και αν τα καταφέρουμε, η αντίδρασή μα σε εξωτερικά προβλήματα και σε κρίσει θα συνδυάζεται με κάποιες κοινέ δράσεις στον τομέα της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάπτυξης. Πιστεύω ότι με ένα τέτοιο συντονισμό θα έχουμε πραγματικά ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Ροτρίγκεθ Πινιέρο από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μίμητσα, εδώ είμαι. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας διαβιβάσω συγγνώμη του Προέδρου της Επιτροπής μας, του κυρίου Μπέντ Λάγκε, δυστυχώς κολλείεται, θα ήθελε να είναι παρόν, αλλά ε, προείσταται στη συνεδρίαση των συντονιστών για την αξιολόγηση της ακρόσης της κυρίας Μάστρομ μου ανέθεσε να σας διαβιβάσω την ερώτηση που συμφωνήθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες της Επιτροπής μας. Όπως γνωρίζετε, το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση για την ανάπτυξη ε, και ε, το εμπόριο για να δώσει νέους προσανατολισμού στην εμπορική πολιτική μετά την οικονομική κρίση. Σε αυτή λοιπόν τη στρατηγική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνε και τη χρηματοοικονομική βοήθεια και τις πολυμερείς ε, εμπορικές προτιμήσεις, κάνοντας μια διαφοροποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και σας ερωτώ, μπορείτε λίγο να μας πείτε ε, αν απέδωσε αυτή η εστίαση, πώς την έχετε αξιολογήσει, εάν αναλάβετε αυτό το χαρτοφυλάκιο, θα συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια και ποια είναι τα νέα μέτρα που θέλετε να υιοθετήσετε για να γεφυρωθεί το χάσμα με τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακόμα και πριν ε, ε, τους στόχους ανάπτυξης, ε, τους βιώσιμους και αιφόρους Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να επανεστιάσει την πολιτική της αυτούς τους στόχους και να την επαναπροσανατολίσει, δίνοντας περισσότερη έμφαση στα θέματα εμπορίου περισσότερο και λιγότερο στα αναπτυξιακά. Τώρα έχουμε στραφεί περισσότερο στους αναπτυξιακούς στόχους, να δούμε δηλαδή πώς το εμπόριο επηρεάζει την ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών και επίσης τις σχέσεις που έχουμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε πραγματικά αναπτύξει μία σχέση εταιρική, ουσιαστική, δηλαδή οι ε, μονομερείς ε, εμπορικές ε, προτιμήσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ και των εκεί συμφωνιών χάνουν όλο και περισσότερο τη σημασία τους και αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από τις γενικές μας εμπορικές συμφωνίες όσο και τις οικονομικές με τις χώρες εταίρους μας. Βεβαίως, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ε, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε ε, αναπτυσσόμενης χώρες, ιδιαίτερα οι λιγότερο αναπτυγμένες είναι και πιο ευάλωτες και πιο ε, εύθραυστες και σε κάποια θέματα έχουμε προτιμησιακή σχέση και παραμένει αυτή, δεν θα καταργηθεί, αλλά πολύ ε, συγκεκριμένα. Εγώ θα προτιμούσα μια πιο συνεκτική προσέγγιση για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες πραγματικά να υποστηριχθούν με τις εμπορικές συμφωνίες. Ε, βοήθεια για το εμπόριο, aid for trade και όχι μόνο κάποιες απαλλαγές από δασμούς και ατέλειες. Ευχαριστώ τις δύο αυτές επιτροπές και προχωρούμε στους υπόλοιπους ε, ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Πρώτος ο κύριος Ρουμπίχ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμένα θα με ενδιαφέρε το εξή, γιατί είμαι και εισηγητή για τον προπολογισμό του 2015. Πώ θα αντιδράσετε στι πληρωμές που δεν έρχονται. Γνωρίζετε πολύ ε, ότι έχουμε αναλάβει πολλέ υποχρεώσει και τώρα δεν υπάρχουν τα χρήματα για την αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν καταβάλλονται οι πληρωμές και έχουν γίνει περικοπές ε, στο διοικητικό κόστος και θα πάνε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, απέτησε 1% ετησίως και συνολικά 4% μέχρι το 2020. Επιπλέον, τι θα κάνετε με αυτές τις περικοπές και ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε εδώ και πιστεύετε ότι αυτό μπορείτε να το αντισταθμίσετε. Γιατί περί πρόκειται, το είπατε και προηγουμένως, στην αναπτυξιακή συνεργασία θέλετε να ενισχύσετε τον ιδιωτικό τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο να έρθουν στο προσκήνιο. Πώς θα το κάνετε αυτό. Ναι. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις πιστώσεις πληρωμών για τα αναπτυξιακά προγράμματα και μέσα είναι πραγματικά τεράστιο. πλησιάζουμε σε μια στιγμή που θα έχουν στερέψει τα κονδύλια για μελλοντικές πληρωμές. Ούτε υποχρεώσεις δεν θα μπορούμε να αναλάβουμε. Και μετά τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο δεν θα έχουμε χρήματα να ανταποκρινόμαστε στις ε, υποχρεώσεις μας για το μέσο αναπτυξιακής βοήθειας. Ξέρω πόσο ανητικό είναι αυτό και τι αντίκτυπο ανητικό μπορεί να έχει και για τους δικαιούχους αλλά και για την αρχή που εφαρμόζει όλα αυτά, ε, που είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά τα έργα. Γενικά για το 2014 φαίνεται ότι ...730 εκατομμύρια ευρώ είναι το κενό διότι ήδη εκκρεμούν περσινές πληρωμές που δεν έχουν καταβληθεί και μεταφέρονται για να αυξηθεί ο όγκος των ε, καθυστερημένων πληρωμών και του χρόνου. Αντίστοιχη κατάσταση θα αντιμετωπίσουμε και τέτοια δυσαναλογία ανάμεσα στην ανάληψη υποχρεώσεων και στις πληρωμές. Που θα έρθουν άλλα ας πούμε 300 εκατομμύρια να προσθεθούν ε, στις καθυστερημένες πληρωμές στα αναπτυξιακά προγράμματα. Πέρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Εμείς κάναμε αυτό που θα έκανε κάθε καλός λογιστής. Καθυστερήσαμε κάποιες πληρωμές, επιλέξαμε κάποιες άλλες, σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Ας πούμε οι πιο φτωχές χώρες να μην ε, είναι σε μειονεκτική θέση και με τις ανάγκες τους Τώρα ε, έχουμε περάσει στην πολιτική δράση, πέρα από τη λογιστική. Δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με τον τροποποιητικό και διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2014 και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2015. Και φτάνοντας στην ενδιάμεση αναθεώρηση, αυτά τα θέματα οπωσδήποτε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινό μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκεράρο Σαλόμ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Μιμίτσα. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε το επόμενο έτος. Θα πρέπει να αποδείξουμε και με έργα ότι βρισκόμαστε στην πρωτοκαθεδρία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση δύο βασικών προκλήσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας, τις κλιματικές αλλαγές και την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων θα πρέπει να ξαναβρούμε τη φόρα που χάσαμε στη διάρκεια της κρίσης και στους δύο τομείς αυτούς και χρειαζόμαστε και νέους πόρους και περισσότερους πόρους. Ερωτώ λοιπόν, είστε διατεθειμένος να πιέσετε τις χώρες ώστε να επιβάλλουν το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ένα τμήμα των φόρων αυτών να αφιερωθεί στην αναπτυξιακή συνεργασία. Είστε έτοιμος επίσης να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Ανάπτυξης, ώστε στη Σύνοδο Κορυφής για την Παγκόσμια Διάσκεψη Χρηματοδότης που θα γίνει του χρόνου στην Αντισαμπέμπα για τα Trust Funds και το Bending και άλλα θέματα που, για τα οποία έχει εκφράσει τη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι ένα σημαντικό στοιχείο ή μάλλον μια σημαντική δυνατότητα για την αύξηση της ε, χρηματοοικονομικής και χρηματοδοτικής δυνατότητας των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις ε, για τον κανονισμό Ευρωπαϊκού Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργούν μια πολύ καλή βάση για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό μου χαρτοφυλάκιο και τις ε, δράσεις για τις οποίες είμαι αρμόδιος, πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να, να περιλάβει όλη τα, να, καλύπτει, να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, γιατί μέχρι στιγμής μόνο 11 κράτη-μέλη έχουν δηλώσει πρόθυμα να εφαρμόσουν τέτοιο φόρο. Θα πρέπει όμως η πρόταση να επεκταθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, το κατά πόσο θα, θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν ε, το 0,7, δηλαδή να υλοποιήσουν τη δέσμευση του να αφιερώσουν το 0,7% του προπολογισμού στην αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό θα το κάνουμε αφενός ε, ε, έχουμε, αυξάνοντας τα έσοδα και φυσικά ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι μια τέτοια δυνατότητα, αλλά και η υπάταξη της φοροαποφυγής είναι μια άλλη δυνατότητα για την αύξηση των προϋπολογισμών. Αν καταφέρουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και να αποφύγουμε ε, κάθε χρόνο να γλιτώνω από τη φορολογία 200 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ένωση, να δηλαδή διαφεύγουν τις φορολογίες, πιστεύω ότι έτσι θα αυξήσουμε το αναπτυξιακό δυναμικό μας την χρηματοδότηση της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Έτσι θα μπορέσουν και οι χώρες αποδέκτες να βελτιώσουν την χρηστή διακυβέρνηση και θα έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας περισσότερους πόρους ώστε να αφιερώσουμε στο συνολικό αναπτυξιακό πακέτο. Σας ευχαριστώ. Κύριος Λούκη, από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ähm, Κύριε υποψήφιε, Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την έκθεση ε, πρωτοβουλίας της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ρόλο του δικαιώματος ιδιοκτησίας για την αηφόρο ανάπτυξη και την ευημερία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η έκθεση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση πρωτοβουλίας. Τώρα εσείς πώς προτίθεστε να αναπτύξετε μια στρατηγική για να προωθήσετε αυτούς τους στόχους και να τους εντάξετε στην αναπτυξιακή πολιτική. Έχετε αντίστοιχο τίτλο, θέλετε να ανοίξετε στον προπολογισμό για να χρηματοδοτείτε τέτοια προγράμματα. Κτηματολόγια και τέτοια χρήση κτήσεις γης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αν ναι, πώς προτίθεστε να το χρηματοδοτήσετε. Διότι είναι δεδομένα τα χρηματοδοτικά προβλήματα που αναφέρατε κι εσείς. Πού θα τα βρείτε αυτά τα χρήματα. Θα καταργήσετε απαλού άλλα αναπτυξιακά έργα και αν ναι, ποια είναι αυτά. ευχαριστώ. Η γενική μου προσέγγιση είναι ότι οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανάπτυξης στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου με θέμα τον προγραμματισμό και τις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λειτουργικό προγραμματισμό συγκεκριμένων προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες θα μεριμνήσουμε ώστε τα σχέδια αυτά, τα προγράμματα αυτά να περιλαμβάνουν και ειδικέ ε, δράσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση και την ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ε, επί της γης ή επί, επί των γεωργικών γεών. Θεωρώ ότι με την προσέγγιση αυτή θα έχουμε μια ευρωπαϊκή συνεισφορά στην οικονομική και χρηματοπιστωτική ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεμονωμένων γεωργών και καλλιεργητών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Δεν θα συμβάλλουμε προκειμένου να ενισχύσουμε την, ή να ε, ενθαρρύνουμε την εφαρμογή γεών, αλλά θα συμβάλλουμε ώστε να διευκρινιστούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Στόχος μας και δράσεις μας θα ακολουθήσουν τους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε όλο όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα, συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να μπορέσουν και οι μικροκαλλιεργητές ή μεμονωμένοι γεωργοί να φτιάξουν στιβαρές ε, οικονομίες και να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση και να συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες ε, εξασφαλίζοντας κάποια δικαιώματα ιδιοκτησίας από τις ε, κυβερνήσεις των χωρών τους ένα από Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση σε σχέση με την ε, αναπτυξιακή πολιτική συνεργασία στην ε, Διατλαντική, δηλαδή συνεργασία με τις ε, ΗΠΑ. Αυτή η εντατική αναπτυξιακή συνεργασία ξεκίνησε στη διάσκεψη κορυφής με τη ΣΥΠΑ στα τέλη του 2009. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορέσατε να εξοικειωθείτε με αυτή τη συνεργασία και πώς θα την αναπτύξετε περισσότερο. Thank you very much. I already spoken in... Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη αναφέρθηκα στην εισήγησή μου σε μια ανάγκη καλύτερου συντονισμού των Ευρωπαίων ε, δωρητών. Δεν μίλησα ακόμα και τόσο για τον ε, συντονιστικό ρόλο που θα πρέπει εμείς να αναπτύξουμε και με άλλους ε, δωρητές και ρίως με τη ΣΥΠΑ. Η διατλαντική, ο μάλλον διατλαντικός συντονισμός των δωρητών θα μπορούσε να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κοινή μας αναπτυξιακή συμβολή στον κόσμο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, καθώς και η ΕΠΑ, μαζί με τις ΕΠΑ, δίνουμε το 80% και πάνω της συνολικής βοήθειας, της αναπτυξιακής βοήθειας. Οπότε, εδώ και καιρό Γνωρίζουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες για καλύτερο συντονισμό θα πρέπει να γίνουν με τη ΣΥΠΑ. Ο συντονισμός λοιπόν αυτός θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος και να βελτιωθεί. Και δεσμεύομαι στο να προωθήσω αυτό το συντονισμό ως πλήρη προτεραιότητα της μελλοντική μου ε, δράσης ε, ως τέταρτη προτεραιότητά μου, γιατί ήδη μιλήσα για τρεις προτεραιότητες, θα είναι λοιπόν στην ατζέντα μου ε, και πάλι θα ήθελα να έχω και τη δική σας συμβολή και να λάβω υπόψη μου τις θέσεις σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγονος από την ομάδα Γκουε και πάλι είναι πίσω σας, κύριε Μίμητσα. Το 2001 τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν να πετύχουν ως το 2015 οκτώ διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους ή στόχους της χιλιετίας όπως ονομάστηκαν. Ωστόσο, στον πιο κρίσιμο τομέα, δηλαδή τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ειδικότερα στην ανάσχεση των απολειών στην βιοπικιλότητα όχι μόνο δεν υπήρξε πρόοδος, αλλά βλέπουμε τις μεν παγκόσμιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα να έχουν αυξηθεί κατά 46% από το 1990 ως σήμερα και ολοένα περισσότερα είδη ζωής να τελούν υπό εξαφάνιση. Δεδομένης της επικείμενης έναρξης διαπραγματεύσεων για το παγκόσμιο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να πάρετε για να μην χαρακτηριστεί τελικά ο 21ος αιώνας ως ερημοζωική περίοδος. Yes, indeed. Όντως, ένα από τα προβλήματα ή τις αποτυχίες του πλαισίου των στόχων της χιλιετίας ή τις παραλήψεις. Είναι αυτό που βλέπουμε με τραγικό τρόπο στην κλιματική αλλαγή, στο περιβάλλον και στη βιοπικιλότητα στον κόσμο. Ακριβώς λοιπόν με τους στόχους της χιλιετίας έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα γιατί κυρίως είχαν επικεντρωθεί στην οικονομική ανάπτυξη, για να το πω έτσι ε, σύντομα. Οπότε, στην διάσκεψη Ρίο συν 20 αναπτύχθηκε αυτή η ιδέα που λέγει ότι θα πρέπει να πούμε πολύ πιο στοχευμένα στην αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη και στους τρεις πυλώνες ε, της αηφόρου ανάπτυξης. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Θα πρέπει τα θέματα αυτά της βιοπικιλότητας ε, και τα περιβαλλοντικά να ενταχθούν πολύ περισσότερο και πιο έντονα στις γενικότερες πολιτικές και στην ατζέντα μας. θα πρέπει να μην χαλαρώσουμε, να διατηρήσουμε αυτή τη συνέργεια και τη συνοχή και ε, την ε, βιωσιμότητα και την αηφορία πάντα ε, κάθε πολιτικής και ανάπτυξης και οικονομικής και κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Με όρους βιοπικιλότητας θα έλεγα πραγματικά ότι πολλά είδη ζωής απειλούνται και γέες και δάση και η ευρωπαϊκή δράση δεν θα πρέπει να υπολείπεται αλλά να είναι ηγετική. Ας πούμε, σε ό,τι αφορά την Άγρια Πανίδα, θα πρέπει εκεί να είμαστε ηγετική δύναμη και όχι ε, να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε, πιστεύω. Η κυρία Χόιμπουχ από τους Πρεσίνους, παρακαλώ η πρωτοβουλία των ε, G8 για μια νέα συμμαχία στην αναπτυξιακή βοήθεια προσβλέπει στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Αφρική με εγχωρίες και ξένες ε, ιδιωτικές επενδύσεις, υποστήριξη αυτών και ανάπτυξη και πρόθεση νέων τεχνολογιών. 60% του πληθυσμού της Αφρικής ε, έχει πολύ μικρό κλήρο και είναι στη γεωργική παραγωγή. Αλλά ε, και πάνω από 70% ε, των ανθρώπων που πεινούν ζουν στην Ήπεθρο. Πρέπει να υποστηριχθούν αηφόρες μέθοδοι γεωργίας για την επιβίωση την ίδια των μικρών γεωργών. Σε πολλά αναπτυξιακά προγράμματα της Ένωσης, των κρατών μελών δηλαδή, είναι προτεραιότητα στη συμμαχία για την ε, επισητιστική ασφάλεια, το G8, θα φροντίσετε αυτές οι επενδύσεις να έχουν αποδέκτες μικρούς αγρότες και μικρές αγρότησες με γεωργικές πρακτικές οικολογικές, όπως ε, λέγει και ο ε, αρμόδιος εισηγητής του ΙΕ για το δικαίωμα την τροφή για να προστατευτούν τα δικαιώματα των μικρών αγροτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε κλήρο. Είπατε μερικά σχετικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και σε πόσιμο είδωρ ή στα δικαιώματα ε, να ε, έχουν ε, πρόσβαση σε πολλαπλασιαστικό υλικό, σπόρους, γιατί παραδοσιακά ο κόσμος ανταλλάσσει τους σπόρους, δεν μπορεί να, έχει βάλει χέρι και η βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως. Η εστίαση στους πιο σημαντικούς τομείς για την αηφόρο ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ένα τμήμα της συνολικής ευρωπαϊκής ε, αναπτυξιακής πολιτικής. ήδη πριν ε, τους ε, στόχους και τη διαπραγμάτευση των στόχων για την ε, φόρο ανάπτυξη και την έγκρισή τους είχαμε αρχίσει να αναθεωρούμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου ε, εξαρτώμεθα πάρα πολύ από την κοινή ε, συνεργασία μας και προγραμματισμό κλαδική και τομεακή με τις χώρες δικαιούχους. Δηλαδή οι χώρες αυτές επιλέγουν οι ίδιες σε ποιους τομείς ε, χρειάζονται και επιθυμούν ε, ε, βιώσιμη αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κράτη-μέλη. Έτσι, συμβαίνει με πολλές χώρες με τις οποίες έχουμε εταιρική σχέση και έχουν επιλέξει τη γεωργία, μια βιώσιμη και αηφόρο γεωργία, αντιμετώπιση του υποσυτισμού, και της έλλειψης τροφίμων ως βασικό στόχο. Όπου υπάρχει λοιπόν αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση και αρκετά ποιοτικά προγράμματα για να μπορούν οι μικρογεωργοί να έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν και την παραγωγικότητά τους και τη συνεισφορά τους στην καταπολέμηση του υποσυτισμού και της στόχιας της χώρας. Οπότε, στη Γεωργία εντάξει. Τώρα στα θέματα της ίδρυυσης και της αποχέτευσης ε, δεν είναι πάντα προτεραιότητα αυτά γιατί οι χώρες επιλέγουν περισσότερο τη Γεωργία. Υπάρχουν όμως και περιφερειακά θεματικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν και θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Καστάλντο από την ε, ομάδα FDD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η διακυβέρνηση είναι ένα σημαντικό μέσο για την βιώσιμη καθολική ανάπτυξη, ιδιαίτερα για περιοχές ευαίσθητες ή καταστάσεις μετά από σειράξεις. Μπορεί να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εταιρικές σχέσεις, όχι μόνο για να μειώσει την ε, διαφθορά, αλλά και για να εφαρμόσει κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες που θα γίνονται σεβαστοί για καλύτερη κοινωνική κοκαταμερισμό του πλούτου ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, σεβασμό δικαιωμάτων, ιδιαίτερα εκείνων των μειονοτήτων, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και οι δικαστικές εξουσίες είναι συχνά καθόδη θέματα στις χώρες εταίρους. Ε, Δηλαδή, πιστεύουμε ότι αυτά τα πολιτικά ζητήματα δεν έχουν πάντοτε γίνει ε, σεβαστά. Η ερεσιμότητα θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί μέσω της ατζέντα για τις αλλαγές. Όμως η πολιτική μας ποτέ δεν έχει διακοπεί, γιατί ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβόταν μη χάσει το κύριο της και την επιρροή της σε σχέση με άλλες δυνάμεις. Πώς θα, εσείς θα κρατήσετε μια ευέλικτη στάση σε αυτό το, θέμα ή η ερεσιμότητα θα είναι προτεραιότητα για σας. Θα σκοπεύετε να εγκαθιδρύσετε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισάγει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δωρητή θα έλεγα αυτή την ε, σχέση, την ερεσιμότητα ε, ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σωστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατική ανάπτυξη και το κράτος δικαίου στις ε, χώρες αποδέκτες ως τμήμα του συνολικού πακέτου βιώσιμης αναπτυξιακής συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες εταίρους. Πραγματικά ηγούμεθα σε αυτόν τον τομέα και ε, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σφυριλατηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή θέση και να μπορεί έτσι πιο εύκολα να προωθηθεί στην διεθνή διάσκεψη των ε, δωρητών. Να προσπαθήσουμε αυτό δηλαδή να το έχουμε ως κοινό στόχο για ολόκληρη την κοινότητα των δωρητών. Τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη δράση όσον, για την αιρεσιμότητα, εγώ θα ακολουθήσω τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στις ε, ισχύουσες συμφωνίες, ιδιαίτερα στη Συμφωνία του Κοτονού, όπου θα πρέπει να είμαστε όντως έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τον πολιτικό διάλογο που το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού, γιατί υπάρχουν ήδη και θετικά παραδείγματα αυτού του πολιτικού διαλόγου, ο οποίος ε, αποδίδει καρπούς και μάλιστα έχει πείσει διάφορες χώρες αποδέκτες να αποσύρουν κάποιες από τις πράξεις τους όπως ας πούμε στην Ουγκάντα και την Νιγηρία για τους ε, ομοφιλόφιλους ή την ε, ε, δουλεία. Θα είναι Λοιπόν, αυτή η προσπάθειά μας πριν να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 86, δηλαδή την αναστολή της εμπορική συμφωνίας, θα έχουμε συμφιζημερείς συζητήσει και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις σωστές θετικές πολιτικές απαντήσεις για να συνεχιστεί η βοήθεια, αλλά όχι μέσω των κυβερνητικών διόδων, αλλά άμεσα προς εκείνους που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια. Ευχαριστώ. Όχι, ο κύριος Γιάνσεν από το σημείο γεγραμμένος, για τρία λεπτά. Ή μάλλον ένα λεπτό, Πρόεδρε, όπως και τα φάρμακα και αναπτυξιακή βοήθεια έχει παρενέργειες που καμιά φορά είναι χειρότερες από το, την ίδια την αρρώστια. Η βοήθεια μπορεί να δημιουργήσει εθισμό και αυτή. Και υπάρχει Επίσης η δυνατότητα ε, λανθασμένης χρήσης του φαρμάκου. Ας πούμε σκάβουν κάτι σύραγγες εκεί και φτιάχνουν και οβίδες ε, τέτοια μέρη που δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς σκέφτεστε, κύριε υποψήφι, να αντιμετωπίσετε αυτές τις παρενέργειες και τις ανεπιθύμητες επίσης επιδράσεις αυτού του φαρμάκου που λέγεται αναπτυξιακή βοήθεια. Uh, Ό,τι κάνουμε στην αναπτυξιακή συνεργασία και στο πλαίσιο αυτό είναι ακριβώς να αποφύγουμε την εξάρτηση, ε, τον εθισμό των ε, δικαιούχων ε, χωρών. Γι' αυτό και εξού προέκυψαν και οι στόχοι και η συμφωνία για την αλλαγή των στόχων για να γίνουν αηφόροι και βιώσιμοι και βασίζεται αυτό σε μια εταιρική σχέση δωρητών και δικαιούχων. Θέλουμε πραγματικά να σπάσει αυτή η περίεργη σχέση που καμιά φορά νοείται και ως φιλανθρωπία. Δεν είναι λιμοσύνη, δεν μας αρέσει αυτή η ιδέα. Θέλουμε να είμαστε εταίροι αναπτυξιακοί για τις αναπτυσσόμενες χώρες από αυτό ε, απαιτεί και τη δική του συνεισφορά και τη δική του προσπάθεια για καλύτερη διαχείριση των ίδιων των πόρων τους. Και καλύτερη παρακολούθηση φυσικά απαιτεί αυτό από πλευράς μας για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Αυτά λοιπόν είναι αλληλένδετα ως διαδικασίες και Έτσι θα αυξήσουμε και την αποτελεσματικότητα για να πιάνουν τόπο τα λεφτά μας. Δεν μας ενδιαφέρει το ποσό, δηλαδή η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Όλο και περισσότερο προς εκεί προσανατολιζόμαστε στα ποιοτικά στοιχεία και στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας αυτής. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα παρακολουθούμε και πολύ στενά μάλιστα εκ του σύνεγγυς και είναι προτεραιότητά μας. Ευχαριστώ. E Η κυρία Ζαμπόρσκα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μίμητσα, σε μία κοινή δήλωση που προσαρτήθηκε στο ε, μέσω αναπτυξιακής συνεργασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 20% το προπολογισμό αυτού του μέσου να αφιερωθεί σε βασικές στοιχειώδεις κοινωνικές υπηρεσίες και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το οριζόντιο ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πρόσφατα όμως, κατά τη διάρκεια του στρατηγικού διαλόγου, ο Επίτροπος Πίμπαξ αναφέρθηκε σε αυτό το 20% λέγοντας ότι προορίζεται στην κοινωνική ένταξη και στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Ε, πρόκειται για μια πολύ ευρύτερη ε, ερμηνεία. Μπορείτε λοιπόν να μας διευκρινίσετε κύριε Επίτροπε πώς ε, θα μεριμνήσετε ώστε το 20% του μέσω αναπτυξιακή συνεργασία να χρησιμοποιηθούν για τι στοιχειώδει κοινωνικέ υπηρεσίε και τη δευτεροβάθμια ε, εκπαίδευση όπω είχε αρχικά προβλεφθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση για το πραγματικό περιεχόμενο του στόχου του 20% για τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες είναι μια συζήτηση που βρίσκεται να εξελίξει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένα της Ειδικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Από την αρχή, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σαφής, ότι το 20% δηλαδή ε, για τις κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να, το 20% αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τις στοιχειώδεις, τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή ήταν από την αρχή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κατά τη γνώμη μου, ο στόχος αυτός ε, είναι υλοποιήσιμος στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου και παρόλο που δεν θα είναι εύκολο να τον υλοποιήσουμε, δεν θα αφιστώ προσπαθειών ώστε να ληφθεί υπόψη το θέμα αυτό και τα αναπτυξιακά κονδύλια να αφιερωθούν κατά 20% στην κάλυψη των στοιχειωδών κοινωνικών υπηρεσιών και της εξασφάλισης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ευχαριστώ ο κύριος ε, Σίλβα Πενέιντα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Περέιρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη μπορεί να σας φανεί περίεργη. Σας ερωτώ λοιπόν, τι είδους επίτροπος φιλοδοξείτε να γίνεται. Γιατί έγινε λόγος για τη συνοχή των πολιτικών απαραίτητος παράγοντας για την ε, επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής. Δεν συμφωνείτε όμως ότι με του, τις διαδικασίες συντονισμού και διατησίες που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειαζόμαστε έναν πολιτικά ισχυρό επίτροπο έτοιμο και πρόθυμο να δώσει τις μάχες του στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής πολιτικής και σας ρωτώ αν είστε αποφασισμένος και έτοιμος να γίνετε τέτοιος πολιτικά ισχυρός και αποφασιστικός επίτροπος. Σε ό,τι αφορά την συνοχή και με τη μεταναστευτική πολιτική. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική αν δεν έχουμε ε, μια πτυχή συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης. Ερωτώ λοιπόν πώς η δική σας αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που θα ευνοεί τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. Σας ευχαριστώ. Μία προσέγγιση συντονισμένων και συνεκτικών πολιτικών όπως πρότεινε και ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, συντονισμός λοιπόν και συνοχή δεν σημαίνει υποτέλεια ε, κάποιων ε, επιτρόπων, των επιτρόπων στους αντιπροέδρους που είναι συντονιστές, γιατί κάθε επίτροπος θα έχει την δυνατότητα να υποβάλει τις προτεραιότητες του και τις προτεραιότητες πολιτικής του και να συμβάλλει σε ένα συντονισμένο επιτυχές αποτέλεσμα. Εγώ θα Ήθελα να είμαι ένας αποφασιστικός ε, άνθρωπος και επίτροπος. Δεν θα δεχτώ αδιαμαρτύρητα πρόταση άλλου αντιπροέδρου ή άλλου επιτρόπου, αλλά παρόλα αυτά είμαι υπέρ του διαλόγου στο σώμα των επιτρόπων για τις πολιτικές και υπέρ του διαλόγου και του συντονισμού στις ε, ομάδες συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτή ε, αυτήν την άποψη έχω ήδη μια καλή εμπειρία, γιατί ως Επίτροπος Αρμόδιος για θέματα κατανάλωσης ε, έπρεπε να συνεργαστώ με άλλους 11 επιτρόπους για να θέσουμε τα συμφέροντα και την προστασία των καταναλωτών ως προτεραιότητα και άλλων πολιτικών και να ληφθούν υπόψη αυτά τα δικαιώματα του καταναλωτή σε όλες τις πολιτικές ένωσες. Με βάση την εμπειρία που αποκόμισε λοιπόν μέχρι στιγμής θεωρώ ότι τέτοιο συντονισμό χρειαζόμαστε και στην αναπτυξιακή πολιτική. Συντονισμό όμως και όχι υπαγωγή του Επιτρόπου σε άλλες πολιτικές, σε άλλους επιτρόπους. Τώρα, για τη μεταναστευτική πολιτική, πώς μπορεί η αναπτυξιακή να συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Φυσικά, θα πρέπει να δούμε την πολιτική εισδοχής μας και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο ορίζεται και πώς ορίζεται η νόμιμη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη συνέχεια θα πρέπει να ενισχύσουμε το δυναμικό των κρατών μελών ώστε να γίνουν ανθεκτικά στις πιέσεις και να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση επιτυχημένων και ανεπτυγμένων κοινωνιών και στις χώρες προέλευσης, χάρη στην αναπτυξιακή μας βοήθεια και πολιτική. Χρειαζόμαστε λοιπόν την αρρωγή και την αναπτυξιακή πολιτική για να ε, μειώσουμε την πίεση της παράτυπης ε, μετανάστευσης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριο Σουλούκη από τους ε, συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ähm, Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που αφορά χώρες μεσαίου εισοδήματος. Τα τελευταία 10-15 χρόνια παγκοσμίω βλέπουμε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και μια σειρά κρατών έχουν βγει από το καθεστώς της κλασικής αναπτυσσόμενης χώρας. 17 συνολικά ε, χώρες αναδύθηκαν και δεν ε, είναι πλήρη δικαιούχοι αναπτυξιακής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν ε, δικαιώματα και αξιώσεις που βαίνουν μειούμενα. Σε αυτές τις χώρες παραμένει όμως πολύ μεγάλη η φτώχεια. Σύμφωνα με μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, 73% των φτωχών αυτού του κόσμου ζουν σε χώρες που ε, ταξινομούνται ως χώρες μεσαίου εισοδήματος. Εάν στο εξής χάσουν τη διμερή τους αναπτυξιακή συνεργασία, πώς θέλετε εσείς να αντιμετωπίσετε. Ε, φτάνει η βοήθεια σε αυτούς τους θύλακες της φτώχειας. Τι θα τους κάνουμε, θα τους αφήσουμε στη μοίρα τους επειδή στατιστικά βγαίνουν οι χώρες από τη βοήθεια. Το έχετε σκεφτεί αυτό και πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Ε, τα κριτήρια διαφοροποίησης έχουν ε, οριστεί από την ατζέντα για την αλλαγή. Ε, υπάρχει η ένευτη τη σταδιακή ε, ανάδυση και μετάβασης των χωρών αυτών από χαμηλού εισοδήματο σε μεσαίο. Και σταματούν ορισμένα διμερεί προγράμματα όντως. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις όπου υπερισχύουν άλλα κριτήρια ή συνυπολογίζονται εκτός από την οικονομική ανάπτυξη. Ε, το εύθραυστο των χωρών, πόσο ευάλωτες είναι, αν χρειάζονται ε, βοήθεια για πιο χρηστή διακυβέρνηση ή να αντιμετωπιστούν τα επίπεδα ανισοτήτων που υπάρχουν μέσα στην ίδια τη χώρα. Κάτ' εξαίρεση λοιπόν τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας παρατείνονται πάντα σε ε, διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πέντε χώρες Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής που παραμένουν. Δηλαδή δεν είναι άσπρο μαύρο η ε, ε, αποχώρηση. Οι χώρες αυτές που βγαίνουν από τη βοήθεια νομίζω είναι περισσότερο σε θέση να αντιμετωπίσουν την ίδια τους τη φτώχεια από τις πιο ευάλωτες ή τις λιγότερο ανεπτυγμένες, τις οποίες στρέφουμε εμείς τη, βοήθειά μας, σε αυτές που έχουν περισσότερο ανάγκη και που μπορούν να γίνουν περισσότερες αλλαγές. Οι χώρες ε, αυτές λοιπόν μεσαίου εισοδήματο είναι επιλέξιμες για τα περιφερειακά προγράμματα και τα άλλα θεματικά επιμέρους προγράμματα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τέτοια προγράμματα και μπαίνουν και στη νέα εταιρική σχέση που οικοδομούμε μια διαφορετική σχέση εταιρικού τύπου με αυτές τις χώρες. Thank you, Mr. Goins, for the ALDE Group. Ευχαριστώ κύριο από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Εγώ θα αναφερθώ στο θέμα της διακυβέρνησης, η διακυβέρνηση της αναπτυξιακής πολιτικής. Βρισκόμαστε την παραμονή μιας πολύ μεγάλης διεθνούς διάσκεψης το ραντεβού δηλαδή για μετά το 2015. Εμεί ανέκαθεν υπερασπιζόμασταν την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ε, απελευθέρωση ε, χρημάτων που είναι ο πρώτον δωρητής στον κόσμο θα πρέπει να είναι παρκώς φιλόδοξη. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν εδώ ποιος είναι ο πρώτος του χορού ε, στο πλαίσιο της Κομισιόν και επίσης αν εσείς είστε ο πρώτος στο χώρο στα διεθνή φόρα η πολιτική δηλαδή η δική μας έχει ένα πρόσωπο εντός και εκτός ένωσης. Είναι η ερώτησή μου και ο φόβος μου ταυτόχρονα. Μήπως μπορείτε εσείς να με καθησυχάσετε. Thank you. Thank you very much. σας ευχαριστώ πολύ. Η έννοια της αναπτυξιακής πολιτικής που είναι προσανατολισμένη στην εκρίζωση τις φτώχειας μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης ε, φέρει μαζί του ε, διάφορα ζητήματα οργάνωσης ε, όσον αφορά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή συντονισμό ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την Κομισιόν, ήδη εξήγησα ότι θα ήθελα να διατηρήσω αυτόν τον ηγετικό ρόλο ε, όσον αφορά τον συντονισμό της βοήθειας των δωρητών από το κράτη-μέλη όχι μόνο δηλαδή όσον αφορά την επίτευξη των ε, δημοσιονομικών στόχων, το 0,7 σε περίοδο ε, την επόμενη, αλλά και όσον αφορά το συντονισμό της συγκεκριμένου προγραμματισμού, δηλαδή βελτίωση του κοινού προγραμματισμού με τα κράτη-μέλη. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική της Κομισιόν εν γέννη, τότε η πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη βρίσκεται στο η πρώτη γραμμή των μέσων εφαρμογής των ε, στόχων μας. Αυτός είναι ο τομέας όπου ο Επίτροπος Ανάπτυξης και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη δεν μπορούν να είναι ο μόνος παίκτη, θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτά τα στοιχεία του συντονισμού όχι μόνο εντός ε, του προγράμματος, ε, μάλλον της ομάδας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, θα πρέπει να περιληφθούν διάφοροι επίτροποι για την ενέργεια, για το περιβάλλον, τις κλιματικές αλλαγές, τη γεωργία. Δηλαδή απαιτείται η προσέγγιση του καλύτερου συντονισμού για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική. Σας ευχαριστώ, κυρία Σάντσες Καλντέντε από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια, όπως και ο προκάτοχός σας είπατε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για, την, ε, για το πρόγραμμα του Blending και μάλιστα ο προκάτοχός σας ανέλαβε τη δέσμευση να συμπληρώσει και να ενισχύσει τη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ό,τι αφορά αυτό το blending. Αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Καμία βελτίωση δεν βλέπουμε. Δεν είχαμε διαφάνεια εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε μεγάλη διαφάνεια και ασάφεια για τα διάφορα σχέδια και προγράμματα blending. Πώς θα βελτιωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος λοιπόν. Θα κάνετε μια ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ενημερώνοντας για τα σχέδια και προγράμματα που βρίσκονται επιτάπητος για να μπορέσει να κάνει το Κοινοβούλιο έλεγχο για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων, την ε, επίπτωσή του και τις ε, επιδράσεις σε σχέση, την κοινωνία, σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών, το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ. Το blending δεν θα έλεγα ότι είναι επιπλέον προαιρετικό, αλλά ένα συμπληρωματικό τρόπος ενίσχυσης ε, των ε, χρηματοπιστωτικών δυνατοτήτων των δωρητών πέραν της επίσημης αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Δεν είναι στόχος μας να αντισταθμίσουμε ή να ενισχύσουμε το blending για να αντισταθμίσουμε την ελλειπή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά το να συνδυάζουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με επιχορηγήσεις ή με δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες ή από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οδηγεί σε μια διαφορετική κατάσταση και ενισχύει το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Συμβολής. Γιατί όταν συμβάλλουμε στην χορήγηση δανείων, προσφέρουμε μεγάλη βοήθεια. δεν θα γινόταν δυνατότητα, δεν θα υπήρχε δυνατότητα καταβολής. Οπότε η μόχλευση αυτού του, του blending είναι τεράστια. Και αυτό που θέλουμε είναι να χορηγηθούν κονδύλια από τράπεζες σε αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα. Και μάλιστα με όρους ε, και επιτόκια που θα βρίσκονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Κάτι τέτοιο βέβαια και συμφωνώ μαζί σας ε, απαιτεί αυστηρές ε, και διεξοδικές ε, διαδικασίες ελέγχου και γι' αυτό δεσμεύομαι να ενισχύσω τον άτυπο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, της διευκόλυνσης του blending. Συνάδελφοι, είμαστε στα μισά των ερωτήσεων. Η κυρία Σαρχεντίνη τώρα έχει το λόγο ξανά με τους Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Το Κοινοβούλιο μας καλείται να συζητήσει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξόριξη μεταλλευμάτων σε χώρες σε σύραξη. Είναι της Επιτροπού Εμπορίου ε, εθελοντικό σύστημα αυτορύθμισης. Εσείς πώς θα βεβαιωθείτε ότι αυτή η πρόταση αυτή έχει ε, που πραγματικά αντίκτυπο και θα αλλάξει την κατάσταση ε, σε κοινότητες που ασχολούνται με την εξόριξη για να σταματήσει αυτή η μάστιγα σε χώρες τύπου τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Πρέπει να το πω αυτό. Η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και της προηγουμένης Επιτρόπου ε, ήταν αρκετά ε, πενιχρή δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό, συνοδευτικά μέτρα. Εγώ ερωτώ πώς θα εξασφαλίσετε την αξιοπιστία αυτού του εγχειρήματο. Αναγνωρίζω τη σημασία να υπάρξει ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη διευκόλυνση ε, του εμπορίου με περισσότερους ε, φυσικούς πόρους να αξιοποιούνται από τα ε, αναπτυσσόμενα κράτη, αλλά αυτό θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τη χρηματοδότηση ανταρτών, παραστρατιωτικών ομάδων μέχρι και τρομοκρατών. Ε, εδώ έχει σημασία αυτή η προσέγγιση και το θέμα της εξόριξης μεταλλευμάτων σε εμπόλεμες ζώνες. Ναι, υπάρχει ένα σύστημα αυτορύθμισης, ε, πιστοποίησης από τις ίδιες τις εταιρείες που εισάγουν ε, ορυκτά. Αυτό το θέμα το συζητάει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και έχει και ρήτρα αναθεώρησης. Δηλαδή μέσα σε μία τριετία από τη θέση σε ισχύ αυτού του εθελουσίου συστήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει, θα αξιολογήσει ε, και θα εκτιμήσει κατά πόσο αποδίδει αυτή η θελοντική προσέγγιση ή τουλάχιστον την αναμενόμενη σημασία και αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ας δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτή την προσέγγιση να αρχίσει να λειτουργεί για να δούμε αν θα αποδώσει στο μέλλον. Επίσης υπάρχει μια ανάγκη Ε, όχι απλώς να αφήσουμε αυτές τις συμφωνίες στα χαρτιά, αλλά να αναγκάσουμε αυτές τις μεγάλες εταιρείες να μπουν σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια. Με πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και να μην περιμένουμε να ολοκληρωθεί η τριετία της εφαρμογής για να αρχίσουμε να μελετάμε και να αναθεωρούμε, αλλά να έχουμε μια συνεχή και διαρκή παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής. from the EFTD. Γκίλ από την EFTT. Η μετανάστευση είναι σίγουρα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και μάλιστα ιδιαίτερα οι συνάδελφοι από τις νότιες χώρες όπως η, Μάλτα βρίσκονται υπό την πίεση και γονατίζουν υπό την πίεση μαζικής μετανάστευσης και ο δήμαρχος του Καλέ ε, επίσης ε, και οι ψηφοφόροι μου είναι ε, οργισμένοι με την κατάσταση αυτή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε παράγοντες και ναύσματα ώστε να μην έχουμε τέτοια έξοδο από τις χώρες προέλευσης. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εμπορικές συμφωνίες ουσιαστικά ε, επέτρεψε την ε, υλοτομία, την ε, άκρατη υλοτομία, την εκμετάλλευση, υπερεκμετάλλευση των ορυκτών, του ορυκτού πλούτου της Αφρικής και την αλληλεία στα χωρικά είδατα της Αφρικής με μια ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των πόρων της Αφρικής. Και μάλιστα ο κ. Γιουνκέρ στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων ζήτησε από εσά μια νέα αρχή. Δέχεστε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην Αφρική κατέστρεψαν τις προϋποθέσεις για μια οικονομική ανάπτυξη και οδήγησαν πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους και ότι η Αφρική αξίζει μια νέα αρχή, νέα προσέγγιση, δίκαιο, εμπόριο και συναφή βοήθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν συμφωνώ με την περιγραφή που μας κάνατε του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιρροής της στην Αφρική, του αντικτύπου της πολιτικής στην Αφρική. Με την Αφρική έχουμε εταιρική σχέση. Μία εταιρική σχέση που μεριμνά για, που μεριμνά για τη σωστή αξιοποίηση των πόρων από τις ίδιες τις αφρικανικές χώρες και όχι από ευρωπαϊκές εταιρείες. Βέβαια, μπορεί να έχουμε και ιστορικά και πρόσφατα κάποια παραδείγματα που δικαιολογούν ίσως ή δικαιώνουν τις δικές σας απόψεις ή τη δική σας περιγραφή για τους ε, λόγους ε, των μεταναστευτικών ροών από την Αφρική προς την Ευρώπη. Αλλά ακόμη ε, και αυτή η περιγραφή δεν ήταν καλά τεκμηρωμένη γιατί Μόνο το 20% της αφρικανικής μετανάστευσης πηγαίνει προς την Ευρώπη. Το 80% της αφρικανικής μετανάστευσης είτε είναι εσωτερική μετακίνηση είτε ε, μετανάστευση στο εσωτερικό της Αφρικανικής Υπήρου. Φυσικά δεν θα ήθελα να υποτιμήσω τον αρνητικό αντίκτυπο της παράτυπης μετανάστευσης και ο ρόλος μου δεν θα είναι να ορθώσω τύχη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να συμβάλλω στην, στην, στον κρέμισμα των τυχών εντός των Αφρικανικών χωρών, ώστε να μπορέσουν οι χώρες αυτές να δημιουργήσουν στιβαρές οικονομίες, αηφόρο ανάπτυξη και να βελτιώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές τους συνθήκες, που αυτές συμβάλλουν σε μια αναγκαστική ουσιαστικά μετανάστευση, γιατί η μετανάστευση για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους ε, είναι μία άνθρωση σχεδόν επιβολή προς τους μετανάστες που δεν έχουν τι άλλο, δεν έχουν άλλη λύση. Και φυσικά θα θέλαμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο της ε, νόμιμης ε, μετανάστευσης στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις στην Αφρική. Κύριε Μίτσα, παρακαλώ, μην Παραδένετε το χρόνο σας, ε, γιατί είπαμε δίλεπτες να είναι οι απαντήσεις στο πόλιο. Ο κύριος ε, Σαλβίνη από τους Ευχαριστώ. Πέρα από το γεγονός ότι με την ανεργία που έχουμε στην Ευρώπη πριν να ασχοληθούμε με την νόμιμη μετανάστευση θα ε, φρόντιζα να μειώσω αυτή την ανεργία, Πάντως είμαι εν γέννη υπέρ των, ναι, ας τους βοηθήσουμε αλλά στα σπίτια τους, αντί να χαλάμε λεφτά σε άχρηστες ε, επιχειρήσεις όπως το Mare Nostrum ή το Frontex, να δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα, να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν εκεί, στις χώρες τους. Πώς όμως σκοπεύετε να δείξετε ότι ε, βοηθάμε αυτές, αυτούς τους ανθρώπους. πούμε, ελεύθερη, Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με το Μαρόκο για τα ψάρια και τα απορροκυπευτικά. Εμείς βοηθάμε με τους ε, δικούς μας Ευρωπαίους πολίτες γιατί φτάνουν φτηνά όλα αυτά τα προϊόντα, όμως οι Γάλλοι, οι Ισπανοί παίρνουν λεφτά ε, για να πηγαίνουν να καλλιεργούν στο Μαρόκο και βλάπτουν τους μικρούς εκεί ε, παραγωγούς. Δηλαδή στην ουσία κοροϊδεύουμε τους βορειοαφρικανούς παραγωγούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αναπτυξιακή μας απάντηση και οι δράσεις μας ε, στόχο έχουν ε, να βοηθήσουν ε, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αποδεκτών. Ας πούμε, όσον αφορά την αλληλευτική συμφωνία, κάναμε δραματικές αλλαγές στην κοινή αλληλευτική μας πολιτική. διευκολύναμε τον Ευρωπαϊκό Στόλο να αλλιεύει στα ύδατα των απτυσσόμενων χωρών με την, ε, ε, ε, με την συνεννόηση ότι θα έπρεπε να βοηθούν στην ανάπτυξη της τοπικής αλληλείας και του, στη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχου της. Το ίδιο ισχύει και για την έννοια της ένταξης του ιδιωτικού τομέα στο αναπτυξιακό πλαίσιο. Και εδώ στόχος μας και συμβολή μας, τα προγράμματά μας, οι επιχειρησιακές μας δράσεις δεν υποστηρίζουν, δεν χρηματοδοτούν, δεν βοηθούν ή διευκολύνουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ώστε να εποφεληθούν από την αναπτυξιακή πολιτική. Δεν θέλουμε να ψυχική μας πολιτική να τους ε, να είναι μια εμπορική προσπάθεια για να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές μεγάλες εταιρείες στις δραστηριότητες τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά κύριο λόγο θα θέλαμε εκείνοι να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των πόρων των αναπτυσσόμενων χωρών να συνεργαστούν με μικρές επιχειρήσεις, με γεωργούς, με αλληλείς εκεί, σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέντα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Για πολλά χρόνια ε, είχαμε σημαντική, σημαντικό, σημαντική συμβολή των πρώτων υλών στις διάφορες εμπόλεμες καταστάσεις στο Κονγκό, στη Βερμανία, στην Κεντρική Αφρική, στην Κολομβία εξαιτίας ε, λαθρεπορείου πρώτων υλών χρηματοδοτούνται ομάδες που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και φυσικά πολλές φορές αυτό γίνεται με συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιριών. Πρόσφατα είχαμε μία νομοθετική έκθεση που στο, θέλουμε, που στόχο έχει να μειώσει το συνδυασμό του, το ε, του εμπορίου και της εξόριξης ορυκτού πλούτου με τη χρηματοδότηση τέτοιων στρατιωτικών ε, δραστηριοτήτων. Πώς ε, θα φροντίσετε ώστε να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, γιατί ε, αναφερθήκατε στην κατάσταση αυτή προηγουμένως. Πώς θα εξασφαλίσετε όμως παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθετικής αυτής έκθεσης και πώς θα ζητήσουμε από τις εταιρείε αυτές να αναλάβουν την ευθύνη τους. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την διαφθορά, την ε, νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες μορφές κατάχρησης των αναπτυξιακών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες ή ε, ίδιους πόρους ε, για την ανάπτυξη, αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής μας δράσης. Και στόχος μας είναι να αποτρέψουμε τέτοιες περιπτώσεις κατάχρησης και διαφθοράς. Και φυσικά έχουμε πολιτικό διάλογο με τις χώρες αυτές και άλλες μορφές συνεργασίας για να ελοπίσουμε αυτό το στόχο. Και φυσικά θα πρέπει το εμπόριο να γίνει πιο βιώσιμο και να διευκολύνουμε τις εμπορικές ροές από τις χώρες αυτές, ώστε να αυξήσουμε και τα έσοδά τους για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να διαρρήξουμε το δεσμό μεταξύ της ε, παράνομης χρήσης ε, ε, των κονδυλίων από παράνομη λοτομία ή λαθρεμπόριο πρώτων υλών, δαμαντιών ή αξιοποίηση των φυσικών πόρων από τις χώρες αυτές. Έχουμε ήδη σχετικές πρωτοβουλίες και έχουμε προγράμματα πολιτικού διαλόγου και ελέγχου της πολιτικής και φροντίζουμε ώστε να υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ των εμπορικών ρυθμίσεων και της παράνομης χρήσης των χρηματοδοτικών κονδυλίων. Και θα συνεχίσουμε στο μέλλον την προσπάθεια αυτή μένοντας συγκεντρωμένοι στο θέμα της παρακολούθησης και της ε, αποτροπής παράνομων δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Κυρία Σλάνη για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υποψήφια Επίτροπε η φοροαποφυγή, η φοροαπάτη και είναι προβλήματα πολύ σημαντικά και παγκόσμια και πρέπει ως τέτοια να αντιμετωπίσουν. Οι φοροαπάτες, φοροαπάτες όμως είναι πολύ ψηλότερες στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι πολυεθνικές πολύ συχνά ε, καταφέρουν να φοροδιαφεύγουν αφαιρώντας έτσι σημαντικούς πόρους. Αντίθετα, η φορολογία είναι πολύ σημαντική πόρο χρηματοδότηση για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα και ποια είναι η δεσμευσή σα προ αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, οι περισσότερε αναπτυσσόμενε χώρε αποκλείονται από τι συζητήσει για τα φορολογικά ζητήματα που γίνονται και τα δημοσιονομικά θέματα που γίνονται στον ΩΣΑ και στο G20. Εσείς ε, συμφωνείτε ότι σε όλες τις χώρες ε, τις στοχές και τις αναπτυσσόμενες ε, θα πρέπει να συμμετέχουν ισομερώς για τον καθορισμό κανόνων και πολιτικών δημοσιονομικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Να, συμφωνώ απόλυτα με τη σημασία που αποδίδεται στα θέματα της φοροαποφυγής και τη τη της δημοσιονομικής με συγχωρείτε, διαχείρισης σε τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και εξίσου σημαντικά εδώ στην Ευρώπη. Όμω, όσον αφορά την αύξηση του δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να είναι πραγματικοί εταίροι και να αναπτύξουν την δική τους εσωτερική ικανότητα να χρηματοδοτήσουν ε, τους ε, αναπτυξιακούς στόχους θα ήμουν υπέρ σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο ΟΗΕ, να τους δοθεί το ίδιο επίπεδο Μάλλον να υπάρχει η ίδια προσέγγιση για να δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες και στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αποτελούν τμήμα αυτών των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων για το πώς θα δημιουργηθεί ένας κοινός μηχανισμός αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής παγκοσμίω. Επίσης ε, βλέπω πως τα προγράμματά μας ε, που βοηθούν στη σωστή διαχείριση, διακυβέρνηση και την οικοδόμηση ε, ικανοτήτων, δυνατοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει όλο ένα και περισσότερο να εστιάζεται σε αυτά τα θέματα της φοροδιαφυγής και της παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας που θα πρέπει να είναι τμήμα συγκεκριμένων δράσεων και του πολιτικού μας διαλόγου αλλά και συγκεκριμένων μέτρων που θα ενσωματωθούν στα προγράμματα που προσφέρουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ κύριος Λούκε. Από την Ίσια έχετε πολλή δουλειά απόψε εσείς. Δύο ερωτήσεις έχω για τομείς πολιτικής, όπου η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον επιζήμια είναι. Πρώτη ερώτηση, εμπορική πολιτική ε, που παραμένουν προστατευμένες γεωργικές αγορές και σε συμφωνίες ελευθερομπορίου. Και η άλλη ερώτηση, εσείς φρονείτε ότι οι γεωργικές αγορές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξουν για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Το δεύτερο, η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων που έχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό εκεί και στα αναπτυσσόμενα κράτη. Θεωρείται σωστό ε, το γεγονός αυτό ότι δανειοδοτεί και χορηγεί ε, προγράμματα αναπτυξιακά και επενδυτικά η τράπεζα ή μήπως αυτό εμποδίζει το να αναπτυχθεί ένα γνήσιο τραπεζικό σύστημα της χώρες αυτή. Γιατί ε, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που παίζει αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών ή την πρόσβαση και τη διάνοιξη των αγορών ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη, αρχίσαμε από τη σύμβαση του ΛΟΜΕ που ήταν μονομερής με το ε, αδασμολόγητο σύστημα πρόσβασης προς την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν ήταν συμβατό με τον ΠΟΕ που αναπτύχθηκε στη συνέχεια. Άρα ε, χρειάστηκε να περάσουμε σε διμερείς συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που θα ανοίξει αυτό πλήρως τις αγορές της Ευρώπης για τα προϊόντα των αναπτυσσομένων χωρών και Τούμπαλιν τις δικές αγορές για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Ανέκαθεν, έχουμε μια αντιμετώπιση ασύμετρη Από πολύ νωρίς ανοίγουν οι ευρωπαϊκές αγορές νωρίς ε, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για τα προϊόντα των χωρών ε, αδεσμολόγητα και χωρίς ποσοστώσεις, ενώ ε, οι χώρες με τη σειρά τους στα πλαίσια της αμοιβαιότητας χρειάζονται κάποιο χρόνο προσαρμογής. Θα το συνεχίσουμε αυτό, αλλά θα πρέπει να βάλουμε μια πιο αναπτυξιακή διάσταση στις συμφωνίες εταιρικής, οικονομικής και εμπορικής σχέσης σε χώρες κυρίως με την Αφρική. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συμφωνούσα ότι είναι καλό να παραμένει ε, παρούσα στα δάνεια που χορηγούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά η, η τράπεζα αυτή είναι επενδυτική, δεν είναι αναπτυξιακή θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένο τρόπο συμμετοχής της σε συγκεκριμένα προγράμματα και έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες. κυρία Παγασάου από το Σουλευθέρους. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας κύριε Μιμίτσα. Μία ε, επίτροπος από την προηγούμενη επιτροπή είπε το 2010 ότι η ασφάλεια είναι, ε, βρίσκεται υποκίνδυνο και μάλιστα το 2013 Είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, 109 θυμάτων και στην Γάζα είχαμε, στη Σιέρα Λεώνα, στη Γινέα, στο Πακιστάν, ε, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων έχασαν τη ζωή τους και όχι μόνο από τον ιό έμπολα. Και επίσης οι φανατικοί τρομοκράτες ενίσχυσαν την κρίσιμη κατάσταση με, με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου για το ανθρωπιστικό προσωπικό. Και μάλιστα ε, από τις πολιτικές που χρηματοδοτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές οργανώσεις μας ζητούν ε, μεγαλύτερη ασφάλεια. Οπότε, πέραν της αποτελεσματικότητας και της συνοχής που φαίνεται ότι σα είναι προσφυλή έννοιες θα πρέπει να μιλήσουμε για θετικά μέτρα και συγκεκριμένα που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των, των, των μελών αυτών των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Επίσης πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τα μέλη τέτοιων οργανώσεων ανθρωπιστικού προσωπικού. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο της ανθρωπιστικής βοήθειας ή ιατρικού προσωπικού ή νοσηλευτών, η ασφάλεια όλων αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα στα λειτουργικά κριτήρια που εφαρμόζουμε κατά τον προγραμματισμό της αναπτυξιακής μας βοήθειας. Της βοήθειας που χορηγούμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέχρι στιγμής ε, η συμβαλόμενοι οργανισμοί ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή τοπικοί φορείς, τοπικές αρχές ή οργανώσεις ε, κρατών μελών λαμβάνουν υπόψη τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα χρησιμοποιούν ως ε, σημεία αναφοράς και ως κατευθυντήριες γραμμές στις δικές τους δράσεις. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρούνται κάποια βασικά κριτήρια σε τέτοιες επιχειρήσεις, βασικά κριτήρια ασφάλειας. Επίσης, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το κόστος εκένωσης τέτοιου προσωπικού οργανώσεων που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα σε περίπτωση που δρούν σε περιοχές όπου υπάρχει κρίση. Πιστεύω ότι έτσι θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των τοπικών φορέων και άλλων οργανώσεων και η δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου. Θέλουμε να τις ενισχύσουμε αυτή την άποψη και γι' αυτό θα προβλέψουμε και συμπληρωματική χρηματοδότηση από πλευράς δωρητών για να καλύψουμε και τις πτυχές αυτές. Ο κύριος Χρυσόγονος από την ΚΟΕ. Κάθετε πίσω σας κύριε Μιμίτσα. Επίτροπε, το μέσο ημερήσιο εισόδημα καθενός ανθρώπου από το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού υπολογίζεται σήμερα πως είναι ίσο με το μέσο ετήσιο εισόδημα του φτωχότερου 57%. 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα και μάλιστα μερικοί από αυτούς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στα κράτη-μέλη που έχουν γίνει θύματα μνημονιακών προγραμμάτων με τη συνενοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα ωστόσο με το προήμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, η Ένωση εδράζεται στις αξίες της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ως Επίτροπος Ανάπτυξης, ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε η αναπτυξιακή πολιτική και οι εξωτερικές δράσεις της Ένωσης να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη κατανομή του παγκόσμιου πλούτου. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι η παγκοσμιότητα, η η καθολικότητα των αηφόρων στόχων ανάπτυξης ή των στόχων αηφόρων ανάπτυξης σημαίνει ότι σκοπός μας είναι να μειωθεί μέχρι και να εκριζωθεί η φτώχεια ε, εξίσου στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες και στην Ευρώπη την ίδια. Αυτή η καθολική προσέγγιση θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και την αρχή της αλληλεγγύης στην οποία εδράζεται η αναπτυξιακή μας πολιτική. Εξάλλου είμαστε δεσμευμένοι και από την αντίστοιχη πρόνοια της συνθήκης που καθοδηγεί και διέπει όλη την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας που έχουμε αναλάβει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα επικεντρώσω πάρα πολύ τις δραστηριότητές μου στην πλήρη εφαρμογή των υφισταμένων κειμένων μας. Δηλαδή, στη συνένεσή μας για την ε, ανάπτυξη, αλλά και την ατζέντα για την αλλαγή, όπου ήδη έχουμε ορίσει σαφή κριτήρια ότι η αναπτυξιακή μας βοήθεια θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένη, ε, που θα πει ότι δεν θα κατευθύνεται σε χώρες που σταδιακά βγαίνουν από αυτό το σύστημα και μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια ε, μόνες τους και να διοχετεύσουμε λοιπόν την ε, αναπτυξιακή βοήθεια σε ένα περιορισμένο αριθμό τομέων στις πιο φτωχές χώρες και στις χώρες που μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εστιάζουμε τη δράση μας και στρεφόμαστε προς την εξάλληψη της στόχιας εκεί που είναι πιο κατάφορη ως φαινόμενο. Ευχαριστώ. κυρία Χάουτολ, τον Πρασίνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντας ε, την ε, ανταλλαγή υπόψεων για την μετανάστευση και την ανάπτυξη, παραμένω ανήσυχη, διότι θυμάμαι την επιστολή ε, που σας έδωσε ο κύριος Γιούνκερ σας ανέθεσε την ανάπτυξη κατάλληλων τρόπων για να διαχειριστούμε τις ε, παράνομες μεταναστευτικές ροές. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να είναι τρόπος για να αδαπανηθεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω απλά ναι ή όχι δεσμεύεστε να μην δαπανίσετε τα χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας στην διαχείριση της ε, των, των ε, μεταναστευτικών. Πολύ λίγα υπόθηκαν δε από τον, ε, για τον κυρίαρχο ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη. Πώς στην πράξη θα τα λάβετε όλα αυτά υπόψη ώστε να προωθήσετε την αναπτυξιακή μας ατζέντα. Μάλιστα. Η αναπτυξιακή πολιτική και η συνεργασία είναι μια πολιτική που θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση των μεταναστευτικών ροών και να ελαφρύνει την πίεση προς την Ευρώπη στην περίπτωσή μας, εφόσον δηλαδή συμβάλλει στην οικοδόμηση οικονομιών και κοινωνιών που θα είναι ευημερείς και ευνοϊκές ώστε οι μετανάστες να μένουν στη χώρα τους και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ίδιας τους της χώρας. Η δική μου αντίληψη είναι ότι η, τα χρήματα της ανάπτυξης, οι δράσεις της ανάπτυξης δεν θα πρέπει να εστιάζουν και να κατευθύνονται άμεσα στο να κατασκευαστούν τύχη έναντι των ε, παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω προηγουμένως όταν ε, μίλησε για την καταστροφή τυχών στις χώρες των μεταναστών. <coughs> Πιστεύω λοιπόν πως η καλύτερη συμβολή της αναπτυξιακής πολιτικής δεν θα ήταν να βοηθήσουμε οικονομικά ή με άλλο τρόπο με μέτρα για την πρόληψη των παράνομων μεταναστευτικών ροών, αλλά η συμβολή της αναπτυξιακής πολιτικής θα είναι να συνεργαστούμε με συντονισμένο και συνεπή τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να, να έχουμε πολλαπλή προσέγγιση Προ τα αναπτυσσόμενα κράτη-μέλη για να παρεμποδίσουμε την παράνομη μετανάστευση και να διευκολύνουμε την νόμιμη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Έχασα το χρόνο μου νομίζω. Ναι, κύριε Μιμίτσα, στο τέλο θα έχετε άλλα πέντε λεπτά για να κλείσετε. Ίσως μπορείτε εκεί να ολοκληρώσετε κάποιες απαντήσεις. Ο κύριο Γκίλ από το EFTD. Σα ευχαριστώ. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η ΕΠΑ, οι Συμφωνίε Οικονομική συνεργασία, δεν είναι τίποτα παραπάνω από οικονομικές ε, συμφωνίες. Ακόμα και ευρωπαϊκές ε, ΜΚΟ τονίζουν πως δεν είναι ισορροπημένες αυτές οι συμφωνίες, επιτρέπουν πρόσβαση στην Ένωση, εκεί όπου δηλαδή μπορούν να κάνουν τάμι και να καταστρέψουν τις, τις τοπικές αγορές. Οι ηθαγενείς ε, δεν έχουν πρόσβαση στην Ένωση για προϊόντα τα οποία παράγουν και πολλούν αλλά επιτρέπεται να στολούν πράγματα που δεν, όχι μόνο δεν παράγουν, αλλά ούτε μπορούν να παράγουν, όπως ας πούμε ηλεκτρονικά προϊόντα με ψηλής τεχνολογίας ή ε, τμήματα ε, δορυφόρων. Πολλές χώρες θα υποχρεωθούν σε άμεση και ε, άμεσο ανταγωνισμό με τις επιδοτούμενους παραγωγούς της Ένωσης. Μπορείτε να σχολιάσετε πόσο είναι δίκαιες αυτές οι συμφωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι συμφωνίε οικονομική συνεργασία, εταιρικέ σχέσεις. αυτέ τι διαπραγματευόμαστε υπό την εντολή που συλλογικά δόθηκε αν, μέσω διπηρεσιακού συντονισμού διαφόρων επιτρόπων που ηγούνται των διαπραγματεύσεων. Ε, σκοπός μου είναι ε, να οικοδομηθούν, μάλλον να ενταχθούν περισσότερες αναπτυξιακές πτυχές ε, στις ε, συμφωνίες αυτού του τύπου. Διότι δεν αρκεί να διαπραγματευτούμε και να συμφωνήσουμε ε, επί των της ε, όσο γίνεται περισσότερο πιο ελεύθερης πρόσβασης για την Ευρώπη, για τα προϊόντα ή τα προϊόντα τα οποία θα μπορούσε να, παράγει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να ε, συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι ο αριθμός των προϊόντων που μπορούν να εξάγουν είναι περιορισμένος λόγω της ε, αδυναμίας παραγωγής ή της ανταπόκρισης στις προδιαγραφές, ε, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι υγειονομικές ε, προδιαγραφές που απαιτεί η ευρωπαϊκή αγορά. Και αυτό δεν ε, μπορεί να διορθωθεί μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη σχέση ανάμεσα στην, στο εμπόριο και την ανάπτυξη. Ε, ε, δεν είμαστε σε κάποια φάση όπου μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες περιοχές που πρέπει να ολοκληρώσουν ακόμα τις διαπραγματεύσεις και σκοπεύω να παίξω το ρόλο συντονιστή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Χιμένες ε, Μπεσερίλα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε κύριε Μίμητσα. Δεδομένου ότι στο μέλλον θα έχουμε εμπλοκή όλων των φορέων στην εφόρα ανάπτυξη και αυτή την άποψη και ο ιδιωτικό τομέα είναι σημαντικό φορέα. Και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με απότερο στόχο την καταπολέμηση τη φτώχεια, τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη κοινωνική δικαιοσύνη στι χώρε αποδέκτε. Οπότε κύριε Επίτροπε, πώς θα προωθήσετε την ε, συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των αναπτυσσομένων χωρών, ώστε να γίνει αποτελεσματική αυτή η συνεργασία και τι πολιτικά μέτρα θα αναλυθούν προκειμένου να αναμειχθούν ε, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και δίνοντας ενάυσματα για συντοπική οικονομία και δίνοντας την ευκαιρία και στις γυναίκες να δραστηριοποιηθούν οικονομικά. Επίσης, σε σχέση με τη μετανάστευση και την συνάφεια μετανάστευσης και ανάπτυξης. Πώς θα χτυπήσετε το πρόβλημα και το κακό στη ρίζα του για να αποφύγουμε τα προβλήματα φτώχειας και τη διασύνδεση φτώχειας, διαφθοράς και τρομοκρατίας που είναι σημαντικές μάστιγες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για το δεύτερο σκέλος ερώτησης, θα ήθελα να πω με κίνδυνο να επαναλάβω τις προηγούμενες απαντήσεις μου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Πάντως ανακεφαλαιώνοντας θα ήθελα να πω ότι το συνολικό πλαίσιο και ο σφαιρικός αντίκτυπος της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και ιδιαίτερα της πολιτικής που εντάσσεται στο πρόγραμμα για τις, ε, των αλλαγών και τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης, θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών. για να αποφύγουμε τις μεταναστευτικές ροές από τις χώρες αυτές. Και αυτή θα είναι η συμβολή, η συνεισφορά της αηφόρου αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε να περιοριστεί η μετανάστευση. Τώρα την πρώτη σας ερώτηση την ξέχασα, το πρώτο σκέλος. Μπορείτε να επαναλάβετε το πρώτο τμήμα της ερώτησης σας παρακαλώ την σχέση και την ε, εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ο ρόλος και η ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντικός στο, στο όλο όραμα που έχουμε για την αναπτυξιακή πολιτική. Και ο ρόλος θα επικεντρωθεί και στη χρηματοδότηση επιθετικών δραστηριοτήτων, δηλαδή ο ρόλος του ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα όταν πηγαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και του ιδιωτικού τομέα στις ίδιες αναπτυσσόμενες χώρες, του εγχώριου, των εγχώριων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Φυσικά θα υποστηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Και θέλουμε φυσικά να σεβαστούμε τους ε, στόχους αηφόρου ανάπτυξης ε, και υπό τον όρο ότι θα γίνουν σεβαστοί αυτοί όροι θα ενισχύσουμε την ε, συμβολή του ιδιωτικού τομέα ο κύριος Φοντζουλίκα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε ε, Επίτροπε, έχω μια ερώτηση για την κλιματική αλλαγή που μας αφορά όλους μας, όπου και να ζούμε, όπου και να βρισκόμαστε. Το έτος 2015 θα είναι σημαντική χρονιά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι της αηφόρου ανάπτυξης θα έρθουν να αντικαταστήσουν τους στόχους χιλιετίας και θα, υπάρξει, και θα υπογραφεί μια νέα παγκόσμια συμφωνία κατά της κλιματικής αλλαγής. Είναι προφανέστατο ότι συνδέονται αυτά τα δύο και ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες περιοχές. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύνδεση αηφόρου ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής να μην τονίζεται ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, στην επιστολή που απίφθινε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στον Επίτροπο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας δεν αναφέρεται πουθενά η αηφόρος αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς εσείς θα εξασφαλίσετε να δοθεί ιδέουσα προσοχή αρκετά νωρίς πριν τις διαπραγματεύσεις και ενόψη αυτών για τους στόχους και πώς θα εξασφαλίσετε ε, επαρκή ε, επιπλέον χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής εκτός του προπολογισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια που είναι ήδη υπερφορτωμένος και τεταμένος. ανεξαρτήτως των όσων αναφέρουν οι επιστολές που μας έχει απευθύνει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι δεδομένη αυτή η σύνδεση, χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς τη συνεργασία των αρμοδίων επιτρόπων και όχι μόνο των δύο, αλλά και για το περιβάλλον και άλλων, ε, δεν γίνεται τίποτα. Βεβαίως, υπό την έννοια αυτή θα υπάρξει και συνεργασία και συντονισμός σε επίπεδο επιτρόπων και αρχηγών των ε, διαφόρων έργων. Οι στόχοι, όπως είπατε, μετά το 2015 συνδέονται απολύτως με την ε, κλιματική αλλαγή και την αντίστοιχη ε, διάσκεψη. Δεν πηγαίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, συγκλίνουν. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ενισχύσουμε τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακουστεί με τον ίδιο τρόπο και στις δύο διαπραγματεύσεις και στις δύο διασκέψεις. Αυτό δεν απαιτεί μόνο εξωτερική δράση και συντονισμό των ε, προγραμμάτων εκεί επιτόπου, αλλά γενικότερη συνεργασία. Επίσης, Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια της διαπραγμάτευσης και σωστά να ε, προετοιμάζουμε αυτές τις σκέψεις. Προσβλέπω λοιπόν σε συνεργασία με τον Επίτροπο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή αλλά και με άλλους επιτρόπους ε, υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό των Διπροέδρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ως τομέας πολιτικής. Mr. Ο κύριος Λούκε. Λοιπόν, για τελευταία φορά παίρνετε σήμερα το λόγο. Θέλω κάτι να ρωτήσω για την αιρεσιμότητα ε, της αναπτυξιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίσατε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έγιναν πολλές ερωτήσεις για τη μετανάστευση, ιδιαίτερα για την παράνομη μετανάστευση. Ε, θεωρείτε σημαντικό να χρησιμοποιήσετε εκεί και την αρισιμότητα Δηλαδή, οι χώρες δικαιούχοι θα πρέπει να καταπολεμούν τις οργανώσεις διακινητών και λαθρεμπόρων και να τις πατάσουν, να ελέγχουν ε, τους ε, δρόμους και τις οδούς διέλευσης. Και επίσης να ελέγξετε την προθυμία τους ε, ε, αν είναι πρόθυμες να δεχθούν ε, ε λάθρο μετανάστες που απελάβουν η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αν δεν είναι σαφής η χώρα καταγωγής τους. Yes, uh, migration. Ναι. Τα, οι μεταναστευτικές ιδιαίτερα οι παράνομες, απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση και απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο από την Ένωση. Θα πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να περιλαμβάνει δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δράσεις των χωρών διέλευσης, καθώς επίσης και των χωρών προέλευσης, η καταγωγής των μεταναστών. Σήμερα οι μεταναστευτικές ροές αυτές δεν ξεκινούν από εσκεμμένες πολιτικές των αναπτυσσομένων χωρών. Μπορεί να είναι αντίδραση απέναντι στην αποτυχημένη διακυβέρνηση ή στην κατάρρευση του κράτους ή στην κακή οικονομική κατάσταση για άλλους λόγους να φεύγουν. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης τα έχουμε συμπεριλάβει όλα. Σε αυτή την προσέγγιση της ανάπτυξης που βασίζεται στα δικαιώματα. Έχουμε πολιτικό διάλογο, έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, την ε, λεγόμενη αιρεσιμότητα που αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Ακόμα και αν συνδέονται με ε, τις χώρες αυτές και ε, τη ρίζα του κακού που οδηγεί στη μετανάστευση. Είναι όμως μια ευρύτερη πολιτική που έχει να κάνει και με συμφωνίες επανεισδοχής, με χώρες ε, προέλευσης ή χώρες διέλευσης. Για να έχει ε, ουσιαστικό αντίκτυπο όλη αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ, κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη σας, ποια πρέπει να είναι η θέση του πολιτισμού στην αναπτυξιακή πολιτική. Uh, Ορισμένοι ισχυρίζονται πως ο πολιτισμός ε, είναι ή θα μπορούσε να είναι ένα παραμελημένο τμήμα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων της. Αλλά εγώ όχι. Όταν μιλάμε για κοινωνική βιωσιμότητα, αυτό ξεπερνά την απλή παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών μπορεί να είναι τμήμα των ε, δράσεών μας που σχετίζονται με την υγεία, τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά όταν ε, πρόκειται για ευρύτερη κοινωνική βιωσιμότητα, αυτή περιλαμβάνει όλα όσα σχετίζονται με την κοινωνική ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των ε, πολιτιστικών δικαιωμάτων και της πολιτιστικής ανάπτυξης. συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των δυνατοτήτων τους να αναπτύξουν την ταυτότητά τους και την εθνοτική τους ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα είμαι μεταξύ όσων θεωρούν τα πολιτιστικά προγράμματα ως τμήμα της βιωσιμότητας των στόχων των αναπτυξιακών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκώσα του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Αξιότιμε ε, υποψήφια επίτροπε, γνωρίζετε ότι για μας ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ, Αφρικής Καραϊβικής Συνενικού. Υπάρχει μια συμφωνία, λεγόμενη Συμφωνία Κοτονού. Το έτος 2020 αυτή λίγη. Και υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ε, πώς θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθείτε ως Επίτροπος, τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτή η συμφωνία Κοτονού να παραταθεί και να μην λήξει. Θα κάνετε συνομιλίες, θα έχετε επαφές σχετικά. Ε, η Συμφωνία του Κοτονού είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα που δείχνει πώς θα, λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η εταιρική σχέση Βορρά-Νότου. Θα εκπνεύσει το 2020. Έχουμε ακόμη μια πενταετία μέχρι τη λήξη της Συμφωνίας του Κοτονού. Αλλά δεν αρκεί αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα για να προετοιμάσουμε το νέο πλαίσιο μετά το κοτονού. Θα πρέπει ήδη από τώρα να αρχίσουμε τις προετοιμασίες. Ήδη από του χρόνου, σε σχετικά πρώιμο στάδιο, θα εγκαινιάσουμε ευρείες διαβουλεύσεις, ε, στις οποίες θα συμμετέχουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας, προκειμένου να σχεδιάσουμε τη νέα προσέγγιση για το πλαίσιο μετά τη Συμφωνία Κοτονού. Είπα στην εισαγωγική μου ομιλία ότι το θέμα δεν είναι αν θα συνεχίσουμε αυτή την εταιρική μας σχέση με τις χώρες ΑΚΕ, ιδιαίτερα με, την, με τις αφρικανικές χώρες. Οπωσδήποτε και θα τη συνεχίσουμε. Είναι απαραίτητη η συνέχιση αυτής της εταιρικής σχέσης, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες γενικές αρχές που θα διέπουν τη νέα συμφωνία και θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της ε, μελλοντικής μας συνεργασίας και πέραν αυτών των γενικών αρχών να έχουμε και ειδικού μηχανισμούς, ειδικά προγράμματα για συγκεκριμένες αφρικανικές χώρες ή για συγκεκριμένες ομάδες ε, χωρών και. Αυτή είναι μια πρωτόλια ιδέα και θα δείξει η έκβαση των διαβουλεύσεων πώς θα διαμορφωθεί τελικά η προσέγγιση μας ε, για τη Συμφωνία του Κοτονού μετά το 2015. Και φυσικά στη διαβούλευση αυτή θα συμμετέχουν και οι χώρες ΑΚΕ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνς από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω το θέμα αυτό της ανανέωσης της Συμφωνίας του Κοτονού. Μίλησατε για τα πλεονεκτήματα της Συμφωνίας, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στις αδυναμίες της. Περιλαμβάνει ένα μηχανισμό διαβουλεύσεων και πιθανή αναστολή ενίσχυση σε περίπτωση κατάφορης παραβίασης ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτή η ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρυσι, όταν ε, η Ουγγάντα και η Νιγηρία ε, εξέταζαν κάποιες νομοθετικές νομοθεσίες κατά, κατά των ομοφιλοφίλων ε, δεν ήταν επαρκής η αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι μια νέα εταιρική σχέση θα πρέπει να έχει μια πιο ρητή και κατηγορηματική πολιτική υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συγκεκριμένε κυρώσεις. Και πώς θα προστατεύσουμε τους ακτιβιτιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές, ε, δεδομένου ότι η προηγούμενη συμφωνία του Κοτονού δεν ε, προάσπισε δεόντως τα δικαιώματα των μειονοτήτων και πώς θα, φροντίσουμε βάσει το άρθρο 21 της συνθήκης ε, της Λισαβόνας να αποφευθούν διακριτικές μεταχειρήσεις και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ, ο Επιτρόπος Μιμίτσα. Κατά τη γνώμη μου, το πλαίσιο για τη νέα συμφωνία Κοτονού μετά το 2015 θα πρέπει να περιλαμβάνει και να ενισχύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θέση της στις ε, εταιρικέ μας σχέσεις με τις αφρικανικές χώρες. Σε μεγάλο βαθμό θα στηριχθώ στην αξιολόγηση των εφισταμένων μηχανισμών ερεσιμότητας και πολιτικού διαλόγου που έχουμε με τις χώρες ΑΚΕ. Θα ήθελα να παραμείνει αυτή η αρεσιμότητα. Πιστεύω ότι μια τέτοια διαδικασία θα μας βοηθήσει να αντιδρούμε πιο έγκαιρα σε περιπτώσεις παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη και η Ουγγάντα και η Νιγηρία είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου είδαμε ότι ο πολιτικός διάλογος απέφερε καρπούς σε ό,τι αφορά την αποτροπή παραβίασης ή την διακοπή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Πάντως ε, θα ήθελα να έχουμε ευρείες διαβουλεύσεις για τη νέα Συμφωνία Κοτουνού και να έρθω και στην Επιτροπή σας για επίσημο διάλογο προκειμένου να συμφωνήσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης της αιρεσιμότητας. Για να συμβάλλει η αιρεσιμότητα σε ουσιαστική αποτροπή της παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικέντρωση των προγραμμάτων βοήθειας σε όσους πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ. Κύριε Στσέλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μίμητσα, Αναλαμβάνεται το χαρτοφυλάκιο αυτό σε ενδιαφέροντες καιρούς του χρόνου, λίγων οι στόχοι της χιλιετίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται σε αυτό γιατί έχει εξαγγείλει ότι είναι το έτος αναπτυξιακής βοήθειας, δηλαδή εστιάζει πάρα πολύ για το 2015 σε αυτό. Πολλοί όμως από τους στόχους που υιοθετήθηκαν το 2000 απέχουν πόρο από την ολοκλήρωσή τους. Άρα ε, υπάρχει πολλή δουλειά. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ε, βοήθεια να βοηθηθούν οι ίδιοι για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους μετά. Στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Και είπατε πολύ σωστά ότι θα πρέπει η βοήθεια να πηγαίνει σε εκείνους που την έχουν ανάγκη. Και δεν είναι οι θύνοντες εκεί τα καθεστώτα, αλλά οι άνθρωποι και οι λαοί. Οι πόλεις μεγαλώνουν συνεχώς, χρειάζεται υγιεινή, χρειάζεται προστασία υγείας και φροντίδα, παιδεία, καλή διοίκηση, αλλά εκεί δημιουργείται και η κοινωνία των πολιτών, στις πόλεις. Έχετε καμιά αστική ατζέντα λοιπόν στην αναπτυξιακή πολιτική, προτίθεστε να υιοθετήσετε ένα αυτό και ένα δεύτερο. Η αναπτυξιακή πολιτική πολύ συχνά είναι θέμα κυβερνήσεων. Είπαμε όμως ότι 70% των ανθρώπων ε, στην Ένωση είναι υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας. Δηλαδή θα πρέπει να τους έχουμε συμπαραστάτες στο πλευρό μας και να είναι και περιφερειακή υπόθεση αυτή, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κεντρικό επίπεδο και η τοπική αυτοδιοίκηση να ενέχεται σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, για την ερώτηση αυτή. Η οργάνωση για ανάπτυξη των πόλεων είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και πολύ κρίσιμο της αηφόρου ακριβώς ανάπτυξης. Η αστιφιλία και η εξάπλωση των πόλεων απειλεί ε, την Ήπεθρο, όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν ξέρω, στην Ευρώπη είναι ίσως λίγο καλύτερα. Ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος ότι στην Ευρώπη καταφέραμε να διαχειριστούμε ε, την αστική ανάπτυξη με συγκεκριμένες δραστηριότητες, όχι μόνο πολεοδομία και δράση σε τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα είμαστε σε θέση, αλλά έχουμε και ανάγκη να βρούμε ένα τρόπο να μεταφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία, τα προγράμματα και τις δράσεις που έχουμε εμπειρία σε αυτά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ πραγματικά προσβλέπω πάρα πολύ ε, στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης για να συμμετέχουν και στην κοινωνία των πολιτών, για να υπάρχει μεγαλύτερη εφορία ε, στις αστικές ή ε, περιαστικές ή στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα στις μεγαλοπόλεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και η δική τους τοπική αυτοδιοίκηση έχει τέτοιες αρμοδιότητες. Θα μπορούσαμε και μόνο συνεργαζόμενοι με τοπική αυτοδιοίκηση να ξεπεράσουμε κάποια από τα εμπόδια, τους κοπέλους ή τις ε, ανακολουθίες ε, που αντιμετωπίζουμε σε κεντρικό επίπεδο λόγω κακής διακυβέρνησης. Πραγματικά υπάρχει έδαφος εκεί, η απάντηση είναι καταφατική. Περισσότερες οργανώσεις κοινωνίας πολιτών και περισσότεροι οτά να συμμετέχουν σε αυτή την ε, προσπάθεια και στα δικά μας προγράμματα. Thank you. Mr. Μανσκούρ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, για τη Συμφωνία του Κοτονού. Διαπιστώνω πως ε, είμαι ο τρίτος ε, συνάδελφος που θέτω την ίδια ερώτηση και χαίρομαι για το ότι ένα τέτοιο θέμα έχει ε, καλέσει τόσο το ενδιαφέρον σας. Ε, μάλιστα είναι η πιο πλήρης ε, εταιρική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Βορρά-Νότου που υπάρχει μέχρι στιγμής. Θα έχετε το βαρύ έργο να διαπραγματευτείτε του χρόνου αυτή τη συμφωνία συνεργασίας Βορρά-Νότου και θα ήθελα να συμπληρώσω με δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, Πώς σκοπεύετε να επανεισάγετε διάφορες ερωτήσεις, διάφορα θέματα τα οποία έμειναν σε κρεμότητα κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του 2010, ας πούμε το θέμα της ε, δημοσιονομικής διακυβέρνησης, της καταπολέμησης ε, των φορολογικών παραδείσεων, την ενίσχυση των ε, ρητρών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θα είναι η μεγάλη μου προτεραιότητα αυτή, διότι πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε και να ξανασκεφτούμε το καλύτερο πλαίσιο για το μέλλον στις σχέσεις μας με τις χώρες ΑΚΕ, ιδιαίτερα με την Αφρική. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα να ασχοληθώ και να έρθω σε επαφή με τον κόσμο, με όσους μάλλον ασχολούνται με την προσέγγιση για το πλαίσιο μετά το κοτονού και να επισκεφθώ κάποιους ε, από τους ε, Αφρικανούς ηγέτες συμπεριλαμβανομένης της έδρα της Αφρικανικής Ένωσης. Και έτσι σκοπεύω να προετοιμαστώ για την δημόσια διαβούλευση που ήδη ανακοίνωσε ότι θα ήθελα να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, ε, όπου οι συμβολές των διαφόρων ε, φορέων θα είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση στο πλαίσιο μετά το κοτονού. Πάντως διαπιστώνουμε ότι η προσέγγιση μας ε, βασικά θα πρέπει να είναι με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοσιονομική διακυβέρνηση, την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων ε, και της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε, πώς δηλαδή θα το φτιάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο μας μετά το κοτονό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόγκα, ΕΛΚ. Πίσω σας είναι η κυρία Μίμητσα, είναι αντιπρόεδρος ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, προτινόμενε Επίτροπε. Η εταιρική σχέση μεταξύ των υπερπόντιων διαμερισμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώθηκε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Έγινε μια εμβάθυνση των σχέσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερε ανάγκε των υπερπόντια διαμερισμάτων. Αλλά το γεγονό ότι τα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, που στόχο έχει την καταπολέμηση τη μεγάλη φτώχεια, ε, αυτό έτυχε, ε, βρέθηκε στο επίκεντρο των επικρίσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να προτείνεται για την περίοδο μετά το 2020 ένα ιδιαίτερο εργαλείο και μηχανισμό για τα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη που θα είναι πιο ελαστικό από το Αναπτυξιακό Ταμείο και θα εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ. Η χρηματοδότηση άλλων αυτών των ε, υπερπόντιων διαμερισμάτων και δαφών είναι τμήμα της γενικότερης συζήτησης για το πώς θα καλύψουμε τις ε, ιδιαίτερες ε, χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Και πρόκειται για μια συζήτηση που κρατάει εδώ και πολύ καιρό. Και ο παρόν κανονισμός προβλέπει ότι ένα τμήμα του Αναπτυξιακού Ταμείου προορίζεται για τη χρηματοδότηση αυτών των υπερπόντιων διαμερισμάτων και εδαφών. Φυσικά, εγώ είμαι πρόθυμος να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Φυσικά χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο ελαστικές και ευέλικτες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις γίνεται. Το 11ο Αναπτυξιακό Ταμείο προέβλεπε κονδύλια για τα υπερπόντια διαμερίσματα και δάφη που έχουν αυξηθεί κατά 12%. Αυτό βέβαια δείχνει ότι δεδομένων των αντίξεων οικονομικών συνθήκων χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία του Αναπτυξιακού Ταμείου στη χρηματοδότηση των υπερπόντιων διαμερισμάτων και δαφών. Δεν χρειάζεται καν να περιμένουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση ή την ε, ανανέωση της Συμφωνίας του Κοτονού μετά το 2015. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό κατά την έναρξη των ε, γενικών διαβουλεύσεων για την προετοιμασία του πλαισίου της επόμενης συμφωνίας Κοτόνου. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε ε, Προτινόμενη Επίτροπε, πολλοί σας ε, ρώτησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης θέματα που ε, έχουν να κάνουν με την ουσιαστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με πραγματικές υπηρεσίες και καταπολέμηση της στόχης. Για να το κάνουν αυτό οι χώρες θα πρέπει να ε, διαχειρίζονται τους φυσικούς τους πόρους με σωστό τρόπο και είναι πολύ ε, υψηλή η διαφθορά. Ένα τρεις δολάρια περίπου εκτιμάται ε, η κατάξη και διασπάθηση κονδυλίων, το ξέπλυμα χρήματος και η κατασπατάληση των πόρων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα εξασφαλίσει η αναπτυξιακή βοήθεια να πηγαίνει στους πραγματικούς δικαιούχους και να εξυπηρετεί τους πραγματικούς σκοπούς. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Πρώτον, στα πλαίσια της οδηγίας για ε, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 28 κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κεντρικό μητρό των πραγματικών δικαιούχων και τελικών αποδεκτών έτσι ώστε να είναι δημόσιο αυτό το Μητρό. Και δεύτερον, θα δεσμευτείτε ότι θα αναπτύξετε την νομοθεσία αυτή που είπατε για τα ορυκτά σε εμπόλεμες ζώνες έτσι ώστε οι εταιρείε να είναι υποχρεωμένες και όχι ε, σε εθελούσια βάση να δηλώνουν την προέλευση και ε, τον προορισμό των χρημάτων τους. Εξάλλου στις ΗΠΑ κάτι τέτοιο προβλέπεται νομίζω. Ευχαριστώ. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλήματος του χρήματος και όλων άλλων των άλλων τρόπων ε, κατάχρησης ή διασπάθησης ε, της ε, χρηματοδότησης και των τόπιων πόρων είναι σημαντικό στοιχείο της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής ανάπτυξης. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Κροατία, που χρειάστηκε να μετασχηματίσει ε, το κράτος, να κάνει τη μετάβαση προς το κράτος δικαίου, την οικοδόμηση δημοκρατικής κοινωνίας και να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να χτίσει ένα καλύτερο δικαστικό σύστημα ε, κατά τη διάρκεια της προενταξιακής προσπάθειας. Ε, τα δύο τρίτα της προσπάθειας είναι μεταρρύθμιση. Χρειάζονται όλα μεταρρύθμιση και οι νοοτροπίες και τα μυαλά του κόσμου. Και αυτή η ε, εμπειρία από την ε, διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδειχθεί πολύτιμη και στην αναπτυξιακή βοήθεια, κατά πολέμηση της διαφθοράς ε, και στη δικαιοσύνη και στη διακυβέρνηση ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα για ε, παρακολούθηση, για λογιστικό έλεγχο, για δυνατότητες που πρέπει να οικοδομηθούν και τελικά κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Σύντομες απαντήσεις για το Δημόσιο Μητρό, το βλέπω θετικά. Να υπάρξει ένα τέτοιο Μητρό όσο γίνεται πιο δημόσιο και όσο γίνεται πιο ευρύ και ε, συνολικό. Και για το νομικά δεσμευτικό της δήλωσης ε, για τα ορυκτά που εξορίζονται σε εμπόλεμες ζώνες. Προς το παρόν όχι. Ας δώσουμε μια ευκαιρία πρώτα στο εθελοντικό σύστημα και βλέπουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, σας θέσαμε πολλές ερωτήσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις σας, τις επιλογές σας. Εγώ θα ήθελα να συζητήσω λίγο μαζί σας τα όσα συνέβησαν τα τελευταία πέντε χρόνια στην πολιτική, αναπτυξική πολιτική, η οποία δεν είναι πολύ όρημη, είναι πρόσφατη και θα ήθελα να γνωρίζω τι θα είχατε κάνει διαφορετικά από τον σημερινό Επίτροπο. Ποιο είναι το πιο αδύναμο σημείο των τελευταίων πέντε ετών και έπειτα μπείτε στη θέση μας ως μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Εσείς τι θα είχατε κάνει διαφορετικά, γιατί και εσείς έχετε εμπειρία κοινοβουλευτική ως μέλος τη δική μας επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Όταν ανατρέξουμε όχι μόνο στα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά στην ευρωπαϊκή δέσμευση, στην αναπτυξιακή συνεργασία εν γέννη, θα έλεγα ότι οι στόχοι της χιλιετίας, όπως θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν, είχαν ε, εστιάσει στην οικονομική ανάπτυξη, για την οικονομική αηφορία των αναπτυσσόμενων χωρών μόνο. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, η γενική μας προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική ήταν ε, περισσότερο δωρητές ή, εν πάση περιπτώσει, δίναμε βοήθεια. Ενεργούσαμε δηλαδή ως δωρητές προς τους αποδέκτες. Η αλλαγή τώρα όμως είναι μπροστά μας. Το να αλλάξουμε δηλαδή από τους στόχους της χιλιετίας σε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, δεν είναι μόνο κάτι το τυπικό, που τυπικές διαπραγματεύσεις και τυπική υιοθέτηση ενός νέου συνόλου κανόνες. Είναι μια πλήρης αλλαγή πολιτικής προς περισσότερη συνέπεια, περισσότερη συνεργασία ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, η θέσπιση καθολικών ε, στόχων και σε αυτό θα ήθελα να συμβάλλω, να έχουμε δηλαδή την Ευρώπη όχι πια ε, ως, έναν ε, δωρητή πληρωτή, αλλά ως συνεργάτη και παράγοντα ανάπτυξης. Και εκεί θα πρέπει να κρατήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην τομέα της ανάπτυξης, όχι μόνο διότι χρηματοδοτούμε το μεγαλύτερο μέρος των αναπτυξιακών αναγκών των χωρών αυτών, αλλά και επειδή αυτό το κάνουμε με πολύ βιώσιμο και καθολικό τρόπο όπου λαμβάνουμε πολλές πτυχές στις προσεγγίσεις μας και αυτό θέλω το να το Ε, συνεχίσουμε και να μην το αλλάξουμε το συγκεκριμένο στοιχείο. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε τους δύο τελευταίους ομιλητές, τον κύριο Φλέκεστάιν, εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Καταλάβατε ότι χρειαζόμαστε ένα πολιτικό επίτροπο που να είναι πρόθυμος στο όνομα της πολιτικής ε, και της συνοχή στην αναπτυξιακή βοήθεια να μπορεί αυτά να τα υπερασπίζεται στο σώμα των επιτρόπων σε οποιαδήποτε πολιτική της Ένωσης που αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλληλίες, διεθνές εμπόριο κτλ. Και εσείς και οι υπηρεσίες της ΔΕΦΚΟ θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και επίσης χρειαζόμαστε κάποιον που να είναι ανεξάρτητος από την ύπατη εκπρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί και να συνεργάζεται μαζί της για να προαγάγει ε, προοδευτικές πολιτικές ανάπτυξης. Μαζί θα πρέπει να κάνετε τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πλαίσιο αναπτυξιακής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παριθμόν ένα στον κόσμο δωρητής και θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη παρουσία στη διεθνή σκηνή. Έχω την εξή απλή ερώτηση και τελευταία από πλευρά μας. Πώς θα εξασφαλίσετε μια πιο ισχυρή και στεναρή φωνή της Ένωσης σε ένα διεθνέ περιβάλλον. Η συνολική προσέγγιση μου που προσπάθησα να σας εξηγήσω καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης ήταν ακριβώς εστιασμένη πάρα πολύ σε αυτά τα σημαντικά στοιχεία που μόλις αναφέρατε κι εσείς. Στην ερώτησή σας. η οποία ερώτηση με φέρνει πάρα πολύ προς τα καταληκτικά μου σχόλια ε, που θα ήθελα να σας καταθέσω. Είναι πολλά τα θέματα που θέλουμε να είμαστε παρόντες. Ε, πολιτικός, επίτροπος, ανεξαρτησία, κεραιότητα, όλα αυτά. Ε, για θέματα αναπτυξιακής βοήθειας συνεργασία με όλες τις άλλες υπηρεσίες και τις πολιτικές και τους άλλους επιτρόπους. Αυτό που θα πρέπει εμείς να κάνουμε στην εξωτερική μας δράση και στις αντίστοιχες υπηρεσίες δεν είναι τόσο πολύ να εργαζόμαστε ε, σε κάθε το κλειστό περιβάλλον, σε ένα σιλό ε, κατακαιρματισμένα και περιχαρακωμένα. Θα πρέπει να είναι εγκάρσια αυτά τα θέματα και της εξωτερικής πολιτικής, ε, ανθρωπιστική βοήθεια, ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν θέλω να υποταχθεί καμία πολιτική σε καμία άλλη, αλλά να υπάρχει μια ισχυρή συνεργασία και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι επίτροποι και να μην εργάζονται σε στεγανά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να εργαστώ και να συνεργαστώ και με την Αντιπρόεδρο και είπα τη εκπρόσωπο. Είχαμε κάποιες πρώτες ε, συνομιλίες και επαφές που εγγράφονται ακριβώς ε, σε αυτό το πλαίσιο που προσπάθησα να σας εξηγήσω. Εγώ δεν πρόκειται να είμαι ένας ε, επίτροπος υποταγής, αλλά συντονισμού και συνοχής. Και πραγματικά είμαι προσιλωμένος πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Κύριε Στίερ, σε εσά ανήκει το προνόμιο είστε ο τελευταίος ομιλητής ε, της βραδιάς. Σας ευχαριστώ. Ε, και η πρώτη ερώτηση ήταν στα κροατικά. Θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο κάνοντας και την τελευταία ερώτηση στα κροατικά. Στη διάρκεια της ακρόασης ε, μιλήσατε για, την, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα επανέρχομαι στους στόχους αηφόρου ανάπτυξης. Έχουμε 16 στόχους. Και δεν αρκεί να μιλούμε μόνο για τη σωστή διακυβέρνηση, χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Το θέμα είναι στις διαπραγματεύσεις θα φροντίσετε να τροποποιήσετε την ισχύουσα διαμόρφωση ή θα προσπαθήσετε στην εφαρμογή, στη φάση της εφαρμογής να υιοθετήσετε μια εφαρμογή που θα στηρίζεται στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αντίθεση με τους στόχους ε, της χιλιετίας, οι στόχοι της αηφόρου ανάπτυξης θα εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Ποιος θα είναι ο ρόλος σας. Πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και του στόχου ε, υπαριθμό 16 στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Η προσέγγιση μου για όλους τους στόχους αηφόρου και του στόχου υπαριθμών 16 που αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να αναφέρεται σε επιμέρους στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης, δηλαδή και στη δημοκρατία, στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κράτος δικαίου. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε το σχέδιο που έχει συγκεκριμένη διατύπωση. Πάντως, στο Συμβούλιο Ανάπτυξης θα φροντίσουμε, θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος του έτους να υιοθετήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε το κείμενο που αναφέρεται στο στόχο αυτό τώρα πώς θα το καταφέρουμε θα φανεί αυτό από την οριστικοποίηση του εγγράφου και δεν ξέρω τι μορφή θα έχει τελικά το τελικό έγγραφο πάντως εγώ ως αρμόδιος επίτροπος για την οτιξική συνεργασία αν με επιβεβαιώσετε φυσικά ως Επίτροπο, θα φροντίσω ώστε τέτοιου είδους στόχοι, δηλαδή η συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, ε, όλοι αυτοί οι στόχοι είναι σημαντικές ε, πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής και θα πρέπει να ληφθούν ε, ε, ε, υπόψη και να αναφέρονται και στα πολιτικά μας έγγραφα και στα επιχειρησιακά μας έγγραφα. Και θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια και Συνεργασία. Και ακόμη και αν δεν προσδιορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα στους, αναπτυξιακούς, στους ε, στόχους υφόρο ανάπτυξης, σίγουρα στην φάση εφαρμογής ελπίζω αλλά και είμαι ότι θα εφαρμοστούν με ακρίβεια. Εμείς θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου. Αν όχι στην γενική διατύπωση των στόχων αηφόρων ανάπτυξης, σίγουρα στις συγκεκριμένες μας δράσεις για αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταία ήταν αυτή η ερώτηση. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να μιλήσετε μέχρι πέντε λεπτά. Αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα, αν Θέλετε να απαντήσετε σε κάτι που δεν προλάβατε προηγουμένως. Έχετε το λόγο μέχρι για πέντε λεπτά μπορείτε. Παρακαλώ. We are over time and I'm afraid. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας και εσείς φαντάζομαι θα είστε κουρασμένοι όσο και εμείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία σύντομα να ε, προσεγγίσουμε κάπως τη συζήτησή μας και τα βασικά σημεία καθώς οδεύουμε προς το τέλος της ακρόασης. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. Παλιές ιδεολογίες τύπου δωρητού δικαιούχου δεν ανήκουν, δεν χωράνε στο νέο πλαίσιο. Θα είναι σημαντικά τα επόμενα χρόνια για να προσαρμόσουμε στις νέες πραγματικότητες ε, μια νέα εταιρική σχέση για ένα καλύτερο κόσμο. Χρειάζεται αλλαγή υποδείγματος από τους σημερινούς στόχους της χιλιετίας προς στόχους αηφόρου ανάπτυξης και είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για καλύτερη καταπολέμηση της ένδυας μέσω της ένταξης οικονομικών, ε, κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων και μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να οικοδομήσουμε με άλλους δωρητές και νέους φορείς που θα μπουν στην ανάπτυξη. Αντίστοιχα, η προετοιμασία για το πλαίσιο μετά το κοτονού μας επιτρέπει να επαναβεβαιώσουμε την στεναρή μας προσήλωση προς χώρες ΑΚΕ και ιδιαίτερα της Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα όφιλε ε, και θα είναι στο κέντρο αυτών των ε, εξελίξεων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και τους εταίρους της παγκοσμίω. Πώς θα ε, διαμορφώσουμε, ε, θα, ε, τι θα σέψουμε την παγκοσμιοποίηση και πώς θα την αξιοποιήσουμε. Αυτή είναι η νέη στόχη μας. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, προσβλέπω πάρα πολύ συνεργασία μαζί σας για αυτές τις προτεραιότητες και παραπέρα θα αντλήσω ε, πολλά διδάγματα από την παρούσα ακρόαση. Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη στην Ευρώπη που αναδεικνύει το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο και είναι προς και των εταίρων μας και των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ και πραγματικά προσβλέπω συνεργασία μαζί σας για αυτό το τόσο σημαντικό ε, θέμα ε, που θα διαμορφώσει και τον κόσμο μας ολόκληρο τον πλανήτη για τις επόμενες δεκαετίες. Um, Ευχαριστούμε κύριε Μιμίτσα. Να θυμίσω τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια. Σύμφωνα με τους κανόνες μας, εμείς τώρα θα συνεδριάσουμε και θα συντάξουμε επιστολή εξολόγησης. Δηλαδή θα γίνει αυτό και κλεισμένο το θύρον. Κυρία Πρόεδρε, μια παράκληση έχω μόνο. Ο, ο, ο κύριος Ρούμπιχ ε, στο Twitter δεχόμαστε πολλά παράπονα ότι δεν παρακολουθούν την ακρόαση και δεν λειτουργεί σωστά το ίντερνετ στο κοινοβούλιο. Παρακαλώ να διορθωθεί για την επόμενη φορά. I heard the same about the ναι. Ναι, υπήρξε ε, ένα μικρό πρόβλημα. Όσοι δεν είστε συντονιστές παρακαλώ να φύγετε από την αίθουσα και θα κάνουμε την αξιολόγηση, θα στείλουμε την επιστολή στους ε, Προέδρους των ε, Επιτροπών και μετά θα ληφθεί απόφαση ε, στην Ολομέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο το βράδυ, 6 ώρα, έχουμε άλλη ακρόαση. Δεν ξέρω γιατί η Επιτροπή μας έχει όλα τα βραδινά ωράρια. Αύριο στις 6 και ευχαριστώ και τους Ιρμηνείς. Θα συνεχίσουμε σε λίγο.